Bitte doch alle Kolleginnen und Kollegen und die Gäste, die Plätze einzunehmen. Παρακαλώ να καθίσετε όλοι και όλες. Έχουμε το σχέδιο ημερησίας διάταξης. Έχω. Έχουμε τις γνωστές γλώσσες αλλά και τα κροατικά αλλά δεν έχουμε εστονικά και μαλτέζικα. Έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών, 25 τοπική πολιτική από το Schleswig-Holstein, που ασχολούνται με τα θέματα της ενέργειας, των μεταφορών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τους ε, χαιρετίζω. και από τον κύριο Παρνιό έχουμε μια ομάδα, μάλλον δεν είναι εδώ από το Schleswig Holstein, αλλά έχουμε 25 μηχανικούς μεταλλι... μεταλλιολόγους εδώ, από τον κύριο Παρνιό. Είσαστε εδώ. Α, πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Και περνάω στο σημείο 16, λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, στο σημείο. Έχουμε 8 συνεργάτες από την ε, Σενεγαλική Εθνοσυνέλευση επίσης. Και έρχομαι στο σημείο 4 και έχουμε αποφασίσει να συζητήσουμε περίπου 30 λεπτά για το θέμα κοινωτικού συστήματος καταχώρησης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών με εισηγήτρια την κυρία Ρωμάνα Γιόρνταν. Α, είναι παρούσα βεβαίως. Σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο σε σχέση με το θέμα αυτό. Παρακαλώ κυρία Γιόρνταν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την μεταφορά ραδιανεργών υλικών. Προκειμένου να έχουμε ένα ομοιόμορφο σύστημα πιστοποίησης για την μεταφορά τέτοιων υλικών. Ε, προς το παρόν ρυθμίζεται ως εξής. Η μεταφορά και η μεταφορή ενεργών υλικών πρέπει προηγουμένως να έχουν μια άδεια, μια ενιαία άδεια, σε κάθε χώρα μέλος. Και τώρα στόχος μας είναι να το αντικαταστήσουμε αυτό από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Εγώ στηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω πως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορά την ε, αδειοδότηση αυτή. Έτσι θα μειώσουμε και την γραφειοκρατία, το διοικητικό άχθος. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει ένα τέτοιο σύστημα να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Διότι αν έχουμε ένα ενιαίο σύστημα αδειοδότησης, το οποίο αναγνωρίζεται αμοιβαίως από όλες τις χώρες μέλη, τότε σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε και κοινά κριτήρια για αυτή την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών. Γι' αυτό και στην γνωμοδότησή μου ακριβώς αυτό προτείνω, να θεσπιστούν ενιαία κριτήρια ώστε να αποφύγουμε αδυναμίες. Το πρώτο που πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε είναι ο πληθυσμός να μην έχει καμία αμφιβολία για το πόσο καλό είναι αυτό το ενιαίο σύστημα το οποίο θα ισχύσει. Κατά δεύτερον, τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός μεταφορέα με τις απαιτήσει του παρόντος κανονισμού. Εφόσον κάποιο δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Πρέπει δηλαδή να σταματούν την δραστηριότητά του οι μεταφορεί μέχρι που να τηρήσουν όλα τα κριτήρια. Και μόνο τότε να μπορούν και πάλι να συνεχίσουν τι δραστηριότητέ του. Επειδή εφόσον πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό σύστημα, πιστεύω ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται. Όχι μόνο δηλαδή οι χώρες ε, όπου κυκλοφορεί ο μεταφορέας αυτός, παντού να γίνει γνωστή η περίπτωσή του. Επίσης πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι προβλήματα και παρατυπίες μπορεί να λάβουν χώρα και όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία διοδότησης. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι με την ε, δυνατότητα μη συμμόρφωσης του μεταφορέα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα και στην ε, αδειοδότηση, δηλαδή στην αρχή η οποία αδειοδοτεί στην κάθε χώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρω στην ε, έκθεσή μου. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και για αυτές τις περιπτώσεις. Για το θέμα είναι να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους μεταφορείς αυτούς. Όλος ο πληθυσμός δηλαδή. Επίτε, όταν μιλάμε για απλοποίηση της ε, ρύθμισης και της νομοθεσίας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία δεν θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Δεν θα ήθελα δηλαδή να αφήσουμε από την άλλη τις προθεσμίες κάπως ασαφείς. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προθεσμίες. Στην γνωμοδότησή μου το λέω. Λέω ποια πρέπει να είναι, ποιες πρέπει να είναι οι προθεσμίες και προτείνω επίσης όσον αφορά την λειτουργία του συστήματος αυτού, η Επιτροπή να αναφέρεται στο Κοινοβούλιο και για πρώτη φορά τρία χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ της νέας αυτής νομοθεσίας και μετά κάθε πέντε χρόνια. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου. Περιμένω τα δικά σας σχόλια τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σκιώδης εισηγητές τώρα. Ο Τόνι Μάρντενς, ο Κρίς Ντέβις τον αντικαθιστά. Συγγνώμη Κρίς, συγγνώμη. Η Λίντα αντικαθιστά τον Μπάβελ πρώτα. Ευχαριστώ. Μου έδωσε μια δήλωση ο συνάδελφο που θα σα την διαβάσω. Ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί είναι ασθενή. Ευχαριστεί την εισηγήτρια για την πρότασή τη. Συμφωνεί με την ε, αιτιολογική δήλωσή τη και προσβλέπει σε περαιτέρω συζητήσει. Ευτυχώ μέχρι σήμερα δεν, είχαν, δεν έχουν υπάρξει ατυχήματα στη μεταφορά διενεργού υλικού. Πρόκειται ωστόσο για κάτι που πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ασφαλής διαδικασία. Με και το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται σαφώς στην νομοθεσία με υψηλά επίπεδα ασφάλειας για την ελαχιστοποίηση ατυχημάτων. Η προστασία των ατόμων από τη τις συνέπειες ε, της μεταφοράς ε, ραδιενεργών ε, υλικών στο περιβάλλον είναι βασική προτεραιότητα και ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύσουμε το ευρύ κοινό από τους κινδύνους της ραδιενέργειας. Κάθε κράτος μέλος πιστεύει και ο δισηγητής μας πρέπει να έχει το δικαίωμα να νομοθετεί να απαγορεύει τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού στο έδαφος του βάσει κανόνων ασφάλειας ή εθνικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Έχει μία ερώτηση προς την Επιτροπή, μάλλον. Η πρόταση αφορά κάθε μεταφορέα που μεταφέρει ραδιενεργό υλικό από τρίτες χώρες στην Ένωση και από την Ένωση σε τρίτες χώρες. Αλλά μόνο ο δικός. Το ερώτημα έχει να κάνει ε, Διανεργό υλικό που μεταφέρεται αεροπορικά ή για τη θαλασσία οδού. Τι γίνεται με αυτό το υλικό. Επίσης, τονίζει ότι χρειάζεται μια υπεύθυνη στρατηγική για την διάθεση του αδιενεργού, των αδιενεργών αποβλήτων. Ευχαριστεί την εισηγήτρια και προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία μαζί της. Ευχαριστώ. Ο Κρις Ντέιβις. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω δήλωση του κύριου Μάντες ε, που θα σας διαβάσω, απουσία του ιδίου. Συνοπτικά, και για να μην φάω χρόνο, καλωσορίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα ενιαίο σύστημα καταχώρησης που θα μειώσει το διοικητικό άχθος και θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας από τους κινδύνους για την υγεία και, την, και θα αποφύγει την διαφορετική ερμηνεία του κανόνα από τα κράτη-μέλη. Καλωσορίζει επίσης την, τις προτάσεις της συγγήτριας για την επιβολή της εφαρμογής μέτρων που εξασφαλίζουν ότι όταν ο μεταφορέας δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του οι αρμόδιες αρχές των κρατομελών θα μπορούν να αναστείλουν την μεταφορά αργού υλικού και καλωσορίζει τις προτάσεις για περισσότερο εναρμονισμένα κριτήρια που υπέβαλε η συγκήτρια. Επίσης έχουμε μια πρόταση επιπλέον να προσθεθεί μια τροπολογία που θα απαιτεί από τα κράτη-μέλη μέλη που καταγράφουν, κρουταχωρών τους μεταφορείς να επανεξετάσουν την διαδικασία αυτή αν δεν υπάρχει πραγματική δυνατότητα αξιολόγηση. Και βεβαίω επενεί την εισηγήτρια για τη δουλειά, υπόσχεται και συνεργασία και καλά θα κάνει, διότι έτσι πρέπει να κάνει. Μισελ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγήτρια για τις προτάσεις της. Το πρόβλημα όμως είναι κάπως μεγαλύτερο από ότι το θέμα απλώ της καταγραφής των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών. Θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη επαγρύπνηση για την πρόληψη των κινδύνων. Πριν από ένα μήνα υπήρξε εκτροχιασμός βαγονιών που μεταφέρανε βαρέλια με ραδιενεργά υλικά στη Γαλλία. Το πρόβλημα είναι λοιπόν το εξής. Πρώτον, <clears throat> μια εναρμόνιση για τα δοχεία τα οποία μεταφορά τα οποία πρέπει να αντέχουν τους, ε, τα χτυπήματα και τις πυρκαγιές. Επίσης πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για, τη στάθμευση των ε, βαγονιών στα, ε, στους σταθμούς. Στη Γαρόνη, στο σταθμό που είχαν γίνει όλα αυτά τα, είχαν έρθει όλα αυτά τα βαγόνια, είχαν σταθμεύσει φάτσα με το σταθμό αναμονής των επιβατών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρχε ένα πρόβλημα, ένα ατύχημα. Για την πληροφόρηση και τη διαφάνεια. Είναι απαραίτητο οι μεταφορείς να έχουν όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα βαρέλια αυτά, με τα ραδιεργά υλικά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να έχει κάνει ενώπιόν του από ε, εξαντλημένα καύσιμα που μεταφέρονται με, το, με συστήματα όπως το κάστο ή χαμηλότερης ραδιενέργειας υλικά που μεταφέρονται σε βαρέλια. Η Greenpeace στο παρελθόν είχε εμποδίσει τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Αν μπορεί να το κάνει η Greenpeace, ίσως μπορεί να το κάνουν και οι τρομοκράτες. Και επομένως δεν έχουμε καμία εξασφάλιση για την ασφάλεια αυτών των μεταφορών. Τέλος, <clears throat> τα θέματα ελέγχου είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας έλεγχος για την ρήπανση που μπορεί να προέρχεται από τα βαγόνια καστόρ. Υπήρξαν προβλήματα στη Γαλλία που μετρήθηκε η ραδιενέργεια για αυτά τα βαγόνια. Ποιο μα λέει ότι δεν υπάρχει καμία ρήπανση που προκαλείται από τι μεταφορέ αυτέ και ποιο έχει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματο. Είναι η Αρεμά, η Αντεέφ ή κάποιο άλλο φορέα ή ο μεταφορέα. Πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν να τύχουν διευκρίνηση μέσα στα πλαίσια αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Γιανακουδάκη. Κυρία Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ. Η ομάδα μου στηρίζει τη γνωμοδότηση είναι ισορροπημένη. Διότι δημιουργεί ένα απλοποιημένο σύστημα για αδειοδότηση, κάτι το οποίο θα είναι καλό για τις επιχειρήσεις, εφόσον θα υπάρχει μία άδεια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι χωριστή σε κάθε χώρα. Ε, Επίση μιλάει για τον έλεγχο από πλευρά των χωρών μελών στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης. Καλό είναι αυτό. Η μόνη μου ανησυχία, και ίσως κάποιος θα μπορούσε να μου το διευκρινίσει αυτό παρακαλώ, εδώ σημειώνω ότι οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου έχουν ετοιμάσει μια έκθεση που περιλαμβάνει ε, μια νομική βάση που δεν είναι ορθή. Κάποιος μπορεί να μου το διευκρινίσει αυτό. Η Επιτροπή μίλησε για τα άρθρα 31 και 32 που αναφέρονται στην ασφάλεια, ενώ οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου μιλούν για την λειτουργία της αγοράς και θέλουν ε, τέτοια νομική βάση. Μπορεί κάποιος να μου το διευκρινίσει αυτό. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι είναι καλή έκθεση και θα συνεργαστούμε με την εισηγήτρια βεβαίως. Η κυρία Γκροστέτ τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην κυρία Τζόρνταν, την εισηγήτρια, η οποία παρουσιάζει μια έκθεση που πιστεύω ότι είναι πολύ καλά ισορροπημένη, γιατί αναφέρεται σε ένα κοινοτικό σύστημα καταχώρησης των μεταφορέων ραδιανεργών υλικών. Έχω όμως κάποιες επιφυλάξεις. Όταν μιλάμε για κριτήρια ασφάλειας που πρέπει να είναι κοινά μεταξύ μας, προσοχή στις αρμοδιότητες της ε, Euratom. Δεν πρέπει να είμαστε σε αντίφαση με αυτά. Οπότε με απασχολεί το θέμα της μεταφοράς κάποιων αρμοδιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό με ενοχλεί. Γι' αυτό και υπάρχουν τροπολογίες με τις οποίες εκφράζω επιφυλάξεις. Είναι οι τροπολογίες 3, 10 και 16. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν ήδη νομοθετικά κείμενα τα οποία αναφέρονται σε αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα η οδηγία 96-79 της Euratom και η 18 του 2008. Νομίζω λοιπόν ότι τόσα αναφέρονται εκεί υπάρχουν και κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε κάποια αντίφαση. Τώρα η τροπολογία, το σημείο 6 μάλλον, μιλάει για ενίσχυση της δυνατότητας που έχει το κράτος μέλος όπου κυκλοφορούν οι μεταφορείς. Νομίζω ότι και αυτό είναι υπερβολικό γιατί κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια πάυση μεταφορών ραδιονεργών υλικών. Έπειτα το σημείο 7 νομίζω ότι είναι περιτό. Για μένα η τροπολογία μάλλον και Αυτή η μεταφορά αρμοδιότητας και αυτή η δυνατότητα που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίζει, εμένα με ενοχλεί. Έχουμε την Euratom, έχουμε και την ανεξαρτησία των ρυθμιστών που αποτελεί μια βασική μας αρχή. Έχω λοιπόν επιφυλάξεις για αυτές τις τροπολογίες της εισηγήτρες. Κατά τα άλλα νομίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι αρκετά ισορροπημένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά μας ενδιαφέρει το θέμα της συνολικής ασφάλειας, λέει ο κύριος Ζέμπερ. Δεν πρέπει να κάνουμε μια ισοπαίδωση προς τα κάτω. Μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφαλείας. Και δεύτερον, υπάρχει πάντα και η ελευθερία επιλογής του ενεργειακού φορέα. Η κάθε χώρα μπορεί να απορρίπτει την χρήση πυρηνικής ενέργειας, αλλά Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική στάση στα θέματα αυτά της μεταφοράς των ραδιενεργών υλικών. Και θυμάμαι ότι είχαμε στη δική μου χώρα μια μεγάλη πολιτική δυσκολία στα θέματα αυτά. Επομένως δεν πρέπει να υποχρεωθεί κανένα κράτος μέλος να κάνει πράγματα τα οποία δεν θέλει, δηλαδή να μην υποχρεωμένο να δέχεται μεταφορά πυρηνικών υλικών από το έδαφος του. Δεν πρέπει επομένως μέσα από την πρόταση αυτή, από την πίσω πόρτα να παρακαυθούν πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να μην, να υπάρξει ε, μια διασταλτική εφαρμογή της ε, ε, ιδέας επικουρικότητας και να υποχρεωθούν ορισμένα κράτη να αποδεχθούν κανόνες για εξασφάλιση ασφαλείας εάν τα κράτη-μέλη αυτά δεν έχουν αποδεχθεί την πυρηνική τεχνολογία. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα μπορούμε εμεί να προστατεύσουμε του πολίτε μα σε περίπτωση ενό ατυχήματο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κατανοήσουμε. Επομένω, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια κοινοτική, μια ενωσιακή ρυθμίση για όλα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι το θέμα τη μεταφορά αεριακών υλικών μπορεί να είναι ένα πολύ, πολύ σοβαρό πρόβλημα στι χώρε μα. Θα ήθελα να αναφερθεί η Κομισιόν για το ερώτημα που έχει να κάνει με το νομικό πλαίσιο τη νομική βάση γιατί μετά πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ και καλημέρα. Καταρχάς να καλωσορίσω την εισήγηση της εισηγήτριας και την υποστήριξη από τους σκιώδεις. Για την απάντησή σας, όντως υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου μια θέση για την αμφισβήτηση της νομικής βάσης του άρθρου 132 εμείς θεωρούμε ότι τούτο ενισχύεται βάση, πέρα, περαιτέρω βάση των κανόνων ασφαλείας τόσο των μεταφορέων όσο και του κοινού. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με την γνωμοδότηση αυτή. Θα εξετάσουμε ωστόσο το θέμα, θα επεξεργαστούμε μια δική μας νομική θέση και θα την παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι τα κοντέινερ δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης. Ο στόχος της ε, οδηγίας είναι μεταφορείς που μεταφέρουν ισότοπα ε, ιατρικού χαρακτήρα από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για παράδειγμα που είναι μεγάλος ο όγκος ε, έχουν υλικό το οποίο ε, τα υπόλοιπα υλικά σχάσεις ε, ατομικά, ατομικής ενέργειας ε, καλύπτονται από άλλες από άλλα νομοθετικά κείμενα που δεν επηρεάζονται ούτε αλλοιώνονται από τον υφιστάμενο από τον παρόντο κανονισμό. Παρακαλώ. Η συγγητρία. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω τώρα τίποτα πέραν αυτό που είπα και εγώ πληροφόρηθηκα για το θέμα αυτό της νομικής βάσης και το εξετάζω ακόμα στο φως αυτών που ελέγχθηκαν από τους σκιώδεις εισηγητές. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να βρούμε κοινό έδαφος. Θέλω όμως να επισημάνω και εγώ ίδια ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με πυρηνικούς σταθμούς. Μιλάμε για την μεταφορά ραδιενεργών υλικών και μόνο. Όλες οι χώρες, ακόμα και αν δεν έχουν πυρηνικούς σταθμούς, χρησιμοποιούν ραδιενεργά υλικά και τα μεταφέρουν στο έδαφος τους. Ακόμα και η Αυστρία έχει ένα ερευνητικό ίδρυμα το οποίο χρησιμοποιεί τα υλικά αυτά, έχει ένα ερευνητικό αντιδραστήρα. Επομένω με τον τρόπο αυτό εμεί δίνουμε μια προσθέμενη αξία. Οι χώρες με πυρηνικού σταθμού έχουν ήδη πολλή εμπειρία στον τομέα αυτό και μπορούν να συμβάλλουν στο να θεσπιστούν τα κατάλληλα πρότυπα. και εγώ προσωπικά δεν βλέπω καμία δυνατότητα να έχουμε ένα κοινό σύστημα χωρίς να υπάρχουν κοινά πρότυπα. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει δυσπιστία και δεν μπορεί παρά μόνο να επιδεινώσει την κατάσταση σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τις αρμοδιότητες τους σε ό,τι αφορά τις ε, ρυθμιστικές αρχές, τις καθονιστικές αρχές στα θέματα αυτά, για να εξασφαλίσουν ότι γίνεται η σωστή εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Για το θέμα τώρα της ευθύνη σε ό,τι αφορά τη μεταφορά αυτών των υλικών, είναι ο μεταφορέας ο οποίος επέχει την ευθύνη. Και αυτό αφορά όλα τα πυρηνικά υλικά τα οποία μεταφέρονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιόρνταν. 11 Απριλίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. 6 Μαΐου θα ψηφίσουμε. Και έχουμε στις 29 Μαΐου, μάλλον 29 Μαΐου έγινε η ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή και το Σεπτέμβριο θα έρθει στην Ολομέλεια. Έχουμε χρόνο λοιπόν για τα θέματα αυτά. Και τώρα πάλι επανέρχομαι ε, χαιρετίζω τους τοπικούς πολιτικούς από το κρατήριο του schleswig Holstein που έχουν έρθει τώρα και περνάμε αμέσως στις ψηφοφορίες και συγκεκριμένες ψηφοφορία σταματήματος του ορολογίου για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πρόκειται για την προσωρινή παρέκκληση από την οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών θερμοκήπιο. Πέτερ Λίζε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει διενεργήσει πολύ καλά τις διαπραγματεύσεις και θέλω να ευχαριστήσω τον Μάτιο Γκρός, ο οποίος είναι ο εισηγητής της Επιτροπής Μεταφορών. Είχαμε αυτή τη διαπραγμάτευση με την Ελλαδική Προεδρία, η οποία στο παρελθόν είχε απορρίψει όλες τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πετύχαμε όμως ορισμένα πράγματα, συγκεκριμένα μια σαφή διευκρίνηση ότι περιμένουμε ορισμένα στοιχεία από την ε, διαπραγμάτευση στα πλαίσια της ΙΚΑΟ. Ελπίζουμε ότι η ΙΚΑΟ το Σεπτέμβριο θα μπορέσει να καταλήξει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει θετικά στοιχεία και για το περιβάλλον αλλά θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητα των ε, αεροπορικών εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε έτοιμοι να τροποποιήσουμε εάν συμβεί αυτό και την νομοθεσία μας. Εάν όμως δεν υπάρξει κανένα αποτέλεσμα, εμείς θα παραμείνουμε πιστοί στο στόχο μα να συμπεριληφθούν και οι αεροπορικέ εταιρείε στην εμπορία εκπομπών. Νομίζω ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Μέχρι τι 13 Απριλίου θα πρέπει να περατωθεί αυτή η διαδικασία γιατί αλλιώ θα έχουμε πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και η σχετική ε, συνδίκη σύμβαση μάλλον εκπνέει τον Απρίλιο. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να διεκπαιρέσουμε αυτό το θέμα και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ πολύ Πέτερ. και θέλω να σε ευχαριστήσω για την υψηλή ποιότητα αυτής της συμφωνίας. Έχουμε μια ψηφοφορία όπου αρκεί η απλή πλειοψηφία θα γίνει ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 49 έναντι 8 κατά ψήφων και καμία ε, αποχή. Συγχαρητήρια στον Πέτερ Λίζε. Ερχόμαστε στην έκθεση Σλούτα. Πρόκειται για την ανακύκλωση των πλοίων. Είναι κάπως πιο μακροσκελής αυτή η ψηφοφορία. Έχουμε 8 συμβιβαστικές τροπολογίες. Έχετε όλοι τις κάρτε. σας. Περνάμε λοιπόν στο θέμα της ανακύκλωσης. Τροπολογία σε 2 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Σε 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία σε 7 στην επόμενη σελίδα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Σε 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πηδάμε μερικές σελίδες και πηγαίνουμε στην 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 150 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Για την 152. Εντάξει. Όχι. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές. Ας δοκιμάσουμε ηλεκτρονικά. 26. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 160 με τροποποίηση προφορική υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 160 με προφορική τροποποίηση άρχεται ψηφίσατε όλοι ψηφίσατε πέρας απορρίπτεται σαφώς 160 χωρίς την τροποφορική τροποποίηση κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 29 μέχρι 32 όλες μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 161 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 162 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Έχει νόημα. Εκπίπτει, εκπίπτει, δεν έχει νόημα. Καλά. Ψηφίζουμε και το δεύτερο τμήμα, αν θέλετε. 162 δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται έτσι κι αλλιώς. Σε τέσσερα συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και τώρα περνάμε περνάμε στη 45 υπέρ. Κατά. 45 υπέρ. 45 λοιπόν σας λέω υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 192 υπέρ κατά αποχές δεν σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος είναι 192 άρχεται Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έλεγχος για την 52. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. Πράγματι. Ό,τι ψηφίσαμε, ψηφίσαμε. Τι να κάνουμε. Δεν έχει νόημα, έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνουμε. Αν δεν δουλεύει το μηχάνημα, εντάξει. Κάνουμε και πάλι έλεγχο στην 53. Ξαναψηφίζουμε. 52, συγγνώμη, 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 31-31 απορρίπτεται. Ίσως πρέπει να λαδώσουμε το μηχάνημα για να δουλεύει καλύτερα, λέει ο πρόεδρος. 190 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 190 έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται σαφώς. 53 ε, υπέρ. Κατά. Δεκτή. 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 195 υπέρ κατά δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. 195 ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος είναι 196. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 197 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 198 υπέρ κατά αποχές δεκτή. «199 υπέρ και 200 κατά Απόχες. Απορρίπτεται. 203. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 204. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 205. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 <clears throat> υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 206 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 58. υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές δεν έχω ψηφίσει αρκετή, κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίσατε. με ευρία πλειοψηφία εγκρίνεται. 61 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 209 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 201 εκπίπτει και αυτή. 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή ερχόμαστε στην 68 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 τσεκ τσεκ τσεκ 69 έλεγχος Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Σαφής η πλειοψηφία υπέρ για την 69. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.17 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές 217 ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 39-33 2-20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.22 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 76 υπέρ. Έλεγχος για την 2.22. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. 76. Παίρνω ψηφο... να ζητώ από τον κύριο Συνέρκα να μου λέει αν ψήφισε ή, ή αν δεν πρόλαβε. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 223 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.20 Έλεγχος, ναι. 2.23, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Με τα τσαρούχια δεκτή, συγγνώμη. 2.26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.27 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.25 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.28 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Κάνουμε έλεγχο για την 80. Ψηφίσατε όλοι. πέρα. Με μεγάλη διαφορά. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.32. 81 έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 85 υπέρ κατά, αποχές δεκτή. 86 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 87 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 88 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 92 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Έλεγχος στο δεύτερο τμήμα της 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.35 υπέρ. Πρέπει να πάμε στην 94 γιατί το πρώτο τμήμα της 92 έχει γίνει δεκτός. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.36 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 95 έως 98 ομού. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 2.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.40 υπέρ 2.39 έλεγχος εφόσον θέλετε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε και ένας δεν ψηφίζει εδώ. Γίνεται δεκτή. 2.40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 104 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Σε 8 συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 117 το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές έλεγχος 117 τμήμα 2 ψηφίσατε όλοι ψηφίσατε πέρας 117 τμήμα 2 πάλι από την αρχή 117 τμήμα 2 ψηφίσατε όλοι κάποιοι δεν ψηφίζουν καθόλου Κλείνω όμως την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 2.52. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα της 1. Υπέρ. Κατά. Δεκτό. Τρίτο τμήμα της 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.58 υπέρ κατά αποχές απο. δεκτή, συγγνώμη. Αιτιολογικές σκέψεις, 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 128 τμήμα 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 128 Εκπίπτουν οι υπόλοιπε. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 131 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 138 υπέρ, κατά, άποχες δεκτή. 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 141 υπέρ κατά αποχές δεκτή 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Λάθος κουμπί. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία και πάλι. Δύο συνάδελφοι δεν συμμετέχουν, τώρα ψηφίσαμε πέρας ψηφοφορίας. 59-3 με 0 αποχές. Ε, δεύτερη ψηφοφορία, νομοθετικό ψήφισμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 60 έναντι 2 κατά. Γίνεται δεκτή. Συγχαρητήρια κύριε Σλούτερ. Και πρέπει τώρα να σας ρωτήσω αν θέλετε ή όχι να γίνουν διαπραγματεύσεις πρώτης ανάγνωσης. Κύριε Σλούτερ. Ευχαριστώ. Οι συμβιβασμοί εγκρίθηκαν ουσιαστικά και οι υπόλοιπε αλλαγές δεν είναι τόσο σημαντικές. Ελπίζω να μπορέσουμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Μην εγκαταλείψετε την αίθουσα έτσι γιατί πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι το 2015 πολλά πλοία θα έχουν παροπληστεί εξαιτίας ε, άλλων νομοθεσιών όσον αφορά το έρμα των ε, πλοίων. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να τελειώσει αυτή η υπόθεση όσο γίνεται πιο γρήγορα, να ολοκληρωθεί. Έχουμε αλλάξει την πρόταση της Επιτροπής, αλλά η αρχική... Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί η αρχική εκδοχή δεν θα λειτουργούσε. Αν λοιπόν έγκαιρα προχωρήσουμε, θα μπορέσει να λειτουργήσει έγκαιρα και να γίνεται όπως πρέπει ο παραπλησμός και η ανακύκλωση των πλοίων. Κυρία Φιέλνα. Ευχαριστώ. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Σλίτερ. Όταν ήρθε η πρόταση από την Επιτροπή ήταν τελείως διαφορετική. Την αλλάξαμε σημαντικά. Γιατί αυτό που πήραμε ήταν η εμφαρμογή της σύμβασης του Χονγκ Κόνγκ. Τώρα ωστόσο δημιουργήσαμε ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για να εξασφαλίσει τους, ε, την υλοποίηση των στόχων της Σύμβασης του Χονγκ Κονγκ. Κάτι ενδιαφέρον στοιχείο. Ε, μισό λεπτό. Ε, Είσαστε στα πλαίσια διαδικαστικής παρέμβασης. Έχουμε ψηφίσει. Αν θέλετε να θέσετε ένα διαδικαστικό ερώτημα, ναι, αλλά δεν κάνουμε συζήτηση πια. Τα έχουμε συζητήσει όλα. Τώρα μόνο για διαδικαστικό θέμα μπορείτε να έχετε το λόγο. Όχι. Κύριε Ντέβις και εσείς για διαδικαστικό θέμα ή όχι. Να ρωτήσω τον εισηγητή ή την Προεδρία. Τι άποψη έχουν. Θέλουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει μαζί μας. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι υποχρεωτικό να το αποφασίσουμε σήμερα. Μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Χρειαζόμαστε μια ειδική πλειοψηφία. Δηλαδή 35 συνάδελφοι πρέπει να ψηφίσουν θετικά. Και το ερώτημα είναι, θέλετε να ψηφίσουμε σήμερα κύριε Σλούτερ, ναι ή όχι. Ναι. Κρίς, ε, συζητώ με τους Ιρλανδούς επί, σε μόνιμη βάση και στο κοινοβούλιο ήταν, ε, μας βοηθήσαν πολύ, το ξέρουν και το έχουν πρόψη τους. Ψηφίζουμε τότε. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα έχουμε εδώ την ε, συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια σήμερα το απόγευμα. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν από την αίθουσα να πάρουν τα πράγματά τους είτε τώρα είτε μετά την το επόμενο θέμα. Γιατί θα αλλάξει τελείω η αίθουσα και πρέπει να πάρετε όλοι τους φακέλους σας. Γιατί θα αλλάξουν οι θέσει των βουλευτών. Πάρτε τα πράγματά σας λοιπόν μετά το τέλος αυτής της συνεδρίασης. Ψηφίζουμε τώρα για να υπάρξει μια εντολή διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε δική πλειοψηφία, 35 βουλευτές. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. Δύο συνάδελφοι δεν ψηφίσανε. Αυτό είναι προσωπική απόφαση του κάθε ενός. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε την εντολή διαπραγματεύσεων. Και παρόλα αυτά θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σλίτερ για την έκθεσή του και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα αντισυλληπτικά χάπια τρίτης και τέταρτης γενιάς στη Γαλλία. Θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψε με τους εκπροσώπους της Επιτροπής και τον Οργανισμό Φαρμάκων, την ΕΜΑ. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Ρέιν και τον κύριο Βοτόν και στον κύριο Ρωτιόν θα δώσω καταρχήν το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Ρωτιόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μου δίνει την ευκαιρία να έρθω και να σας ενημερώσω σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τα αντισυλληπτικά τρίτης τέταρτης γενιάς και συγκεκριμένα τον Διάνα. Πρόκειται για συνδυασμένα αντισυλληπτικά που περιλαμβάνουν δύο ειδών ε, ε, ορμόνες και τα οποία συνδέονται με ε, προβλήματα εμβολής των ανθρώπων που τα παίρνουν. Έχουν γίνει μελέτες λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε ε, διάφορα στοιχεία, οπότε οι ρυθμιστικές αρχές αποφάσισαν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να ενημερωθεί η πληροφόρηση που δίνεται για τα όργανα αυτά. Ο πρόεδρος της πράκτης ε, Επιτροπής δηλαδή Αξιολόγησης Κινδύνου Φαρμακοεπαγρύπνησης έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής και θα ασχοληθεί με αλλά και τα ωφέλη των συνδυασμένων αυτών αντισυλληπτικών όπως είναι το Ντιάν και θα εξετάσει τις απαντήσεις που έχουν δώσει οι ρυθμιστικές αρχές όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να ενημερωθείτε κι εσείς για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά τις αποφάσεις της Επιτροπής μάλλον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέιν για την πρόσκλησή σας. Εγώ θα σας παρουσιάσω Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η γνώση που έχουμε για τα ωφέλη και τους κινδύνους από τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά και στη συνέχεια θα πω δύο λόγια για το Διάνο. Υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία έχουν εκτιμήσει οι ρυθμιστές και έτσι έχουν ενημερωθεί και τα συμπεράσματά μας. Έπειτα θα αναφερθώ και στα μέτρα για την ε, άμβλεση των κινδύνων. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά όταν χρησιμοποιούνται ορθά ε, έχουν καλά αποτελέσματα για την αποφυγή ανεπιθύμητων ε, ε, εγκυμονήσεων. Στη συνέχεια έχουμε εξαλλογήσει και τους κινδύνους και έχει εξολογηθεί η μείωση των κινδύνων εξομήτριων. Οι επιδημολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι δεν έχουν αυξηθεί κίνδυνοι σε καρκίνων ούτε σε εθνισμότητα. Υπάρχει μια μεγάλη μελέτη η οποία έχει δείξει ότι όσοι χρησιμοποιούν τα ε, αντισυλληπτικά αυτά έχουν μειωμένη πιθανότητες ε, ε, κινδύνου νωρίς θανάτου. Η κίνδυνοι επίσης θρομβώσεων τώρα. Υπάρχει βέβαια ε, κίνδυνος για τις γυναίκες που δεν είναι σε αντισυλληπτικά. Η περίπτωση να υπάρξουν θρομβώσεις από τη χρήση τέτοιων αντισυλληπτικών επίσης είναι πάρα πολύ μικρή. Μόνο μία το χρόνο φαίνεται να έχει τέτοια προβλήματα θρόμβωσης. Μία στις 10.000. Τα αντισληπτικά τρίτης και τέταρτης γενιάς συνδέονται πάντως με την αύξηση κινδύνου θρόμβωσης. Δύο φορές παραπάνω από ότι όσες παίρνουν ε, αντισληπτικά δεύτερης γενιάς. Δύο λοιπόν στις 10.000. Αν λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία από την αρχή της αξιολόγησης, το φέλη πάντως των συνδυασμένων αντισυλληπτικών είναι πολύ παραπάνω από τους κινδύνους. Τώρα, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το τσεπτικό Διάν. Το συνθετικό τους έχει ωφέλη όταν υπάρχουν υπερβολικά ανδρογενή. Οπότε βοηθάει την καταπολέμηση της ακμής, για παράδειγμα. Εφόσον, ε, μάλλον ε, διαφέρει η άδεια για την κυκλοφορία του τσιλεπτικού αυτού από χώρα σε χώρα. Έχει συγχρόνως και αντισυλληπτικό όφελος αλλά δεν δίνεται γι' αυτό το σκοπό. Η αξιολόγηση κινδύνου είναι γνωστή, τα αποτελέσματά της δηλαδή, και αντιμετωπίζεται στην συνταγολόγηση από όλους τους γιατρούς. Πώς λοιπόν το σύστημα έχει αντιδράσει τώρα στα νέα στοιχεία που έχουμε όσον αφορά τους κινδύνους για θρόμβωση από τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά. Ο ρόλος του ρυθμιστικού σώματος είναι να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος, αξιολογώντας όλα τα νέα στοιχεία που έχουμε και βάζοντας στη ζυγαριά το φέλη και τους κινδύνους από τέτοια προϊόντα και να ληφθούν και μέτρα δηλαδή για τον περιορισμό των κινδύνων. Θα σας πω λοιπόν ποια είναι τα κύρια στοιχεία. Πρώτο, 2009 η, η Αρμόδια Επιτροπή για νέα τέτοια προϊόντα έκανε συστάσεις μετά από την ανάλυση που είχε γίνει για τον κίνδυνο θρόμβωσης από αντισληπτικά τρίτης γενιάς, συνδυασμένα. Και το 2009 έγινε μία μελέτη, δημοσιεύτηκε μάλλον μία μελέτη, η οποία επιβεβαίωσε τα προηγούμενα συμπεράσματα. Και πιο πρόσφατα το 2011 μια πιο νέα επιδημολογική μελέτη αναφέρθηκε στους κινδύνους θρόμβωσης από τα αντισλεπτικά τέταρτης γενιάς. Η... Επιτροπή Ευρωπαϊκή για τέτοια προϊόντα πάντως επίσης έφερε νέα στοιχεία και αναφέρθηκε στον κίνδυνο από αντισυλληπτικά ή συναφή προϊόντα τρίτης και τέταρτης γενιάς. Στη συνέχεια είχαμε νέα στοιχεία από τη Δανία και τις Ηνωμένε Πολιτείε που ευθυγραμμίζονται με την θέση της Επιτροπής Φαρμακοεπαγνύπνησης. Στη συνέχεια είχαμε και νέα στοιχεία όσον αφορά τους κινδύνους θρόμβωσης από αντισυλληπτικά που δεν παίρνονται από το στόμα, πάτσες ή άλλα τέτοια. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει αναλύσει η Επιτροπή Αξιολόγηση Κινδύνου Φαρμακοπαγνύπνησης. Το σύστημα πάντως ρύθμισης δεν έχει αντιδράσει μόνο, αλλά φρόντισε να δημοσιεύσει πληροφορίες και προληπτικά μέσω μιας μελέτης που έγινε στις κάτω χώρες, την, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, Γαλλία και Γερμανία. Όλες αυτές οι νέες ε, πληροφορίες λαμβάνονται υπόψη στην αναθεωρωμένη έκθεση. Ποια είναι τώρα τα μέτρα προκειμένου να βληθούν οι κίνδυνοι από θρόμβωση. Το κύριο μέτρο έχει να κάνει με ε, σαφείς πληροφορίες, με καλή ενημέρωση των ε, ιατρών και γενικά του ιατρικού προσωπικού, προκειμένου όταν συνταγογραφεί κάποιο γιατρός τέτοια φάρμακα να γνωρίζει πολύ καλά περί τίνο πρόκειται. Έπειτα υπάρχουν και διάφορα ε, διάφορες πληροφορίες που δίνονται στους ενδιαφερόμενους με φυλάδια. Πέρα λοιπόν από τα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, η... το αποτέλεσμα ανάμεσα ε, της αξιολόγησης ε, κινδύνου και όφελους κλείνει προ όφελο. Βέβαια η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο ελέγχει συνεχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι στοιχεία υπάρχουν για τον κίνδυνο θρομβώσεων αξιολογούνται μόλις ε, λαμβάνουμε γνώση αυτών. Δίνονται επίσης συμβουλέ για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπάρχουν και δελτία ενημέρωση προ του ασθενεί, ώστε να μπορούν να αποφασίζουν έχοντας γνώση των στοιχείων που διαθέτουμε. Αυτό ισχύει και για τους γιατρούς και για τους ασθενείς. Όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλα τα αποτελέσματα των μελετών μας ε, δημοσιεύονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για να κλείσω. κάποια στοιχεία για την ε, επισκόπηση που γίνεται. Έχουμε δύο έρευνες οι οποίες τρέχουν παράλληλα. Η μία είναι για τα συνδυασμένα ορμονικά αντισυλληπτικά που ξεκίνησε το Φεβρουάριο αυτού του έτους μετά από την αίτηση του γαλλικού φορέα για μία σειρά από αντισυλληπτικά συνδυασμένων ορμονών γιατί υπήρχε εντύπωση ότι ήταν αρνητικό το αποτέλεσμα τους σε επίπεδο κόστος ωφέλους για την πρώτη γραμμή και θα έπρεπε να παραμείνει μόνο σε δεύτερη γραμμή, δηλαδή μη ε, αποζημιούμενα φάρμακα. Μετά από όλα αυτά, το φορέας μας έχει αποφασίσει να διευρύνει το περιθώριο αυτής της έρευνας γιατί υπήρχαν και άλλες φαρμακευτικές μορφές όπως patch τα οποία δεν χρησιμοποιούνται δεν περιλαμβάνουν αυτή τη στιγμή στην εμβέλεια αυτής της αίτησης. Συνεχίζουμε λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τα ερώτηματα τα οποία έχουν τέθει από όλες τις φαρμακευτικές και περιμένουμε να πάρουμε τις πληροφορίες αυτές. Άλλες πληροφορίες επίσης θα ληφθούν υπόψη και είναι σημαντικό αυτή η έρευνα η οποία θα γίνει από τον Οργανισμό Φαρμάκων. Δεν θα βασιστεί μονάχα σε αυτά τα οποία μας δίνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και από άλλους φορείς. Θα έχουμε τα αποτελέσματα διαθέσιμα <clears throat> από πέντε μελέτες οι οποίες από δύο μελέτες χρήσης των φαρμάκων αυτών που θα γίνουν σε πέντε κράτη-μέλη και τα οποία θα δώσουν ένα πληθυσμό συνολικά που θα περιλαμβάνεται σε αυτές τις μελέτες που είναι σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε λοιπόν αυτά τα σημαντικά στοιχεία. Και επιπλέον εξετάζουμε και την βάση δεδομένων μας. Έχουμε μια βάση δεδομένων για όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 3,9 εκατομμύρια εκθέσεις. Επομένως θα έχουμε στοιχεία για τα αντισυλληπτικά συνδυασμένων ορμονών. Επιπλέον θα κάνουμε και μία έρευνα όλων των επιστημονικών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε σχέση με αυτό το θέμα. Και επίσης έχουμε ζητήσει να υπάρξει πληροφορία από 220 εταίρους στην νανσεπ που είναι μια πρωτοβουλία μας το Ευρωπαϊκό ε, Δίκτυο των Κέντρων Φαρμακοεπαγρύπνησης και Επιδημιολογίας. Πρόκειται για ακαδημαϊκούς φορείς οι οποίοι κάνουν μελέτες στον τομέα αυτό και τους ρωτήσαμε αν έχουν να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες σε σχέση με αυτά και ερευνητικά πορίσματα. <clears throat> Προβλέπουμε να τελειώσει η συζήτηση τον Ιούλιο εφέτος πριν από αυτή τη συνάντηση θα κάνουμε μια ομάδα ad hoc εμπειρογνωμόνων, εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορούν να πληροφορήσουν την Επιτροπή μας για τα θέματα αυτά. Εφόσον αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθεί την ε, επισκόπηση από την Επιτροπή ΚΡΑΚ και περιλαμβάνει διάφορα ε, ευαίσθητα προϊόντα, θα πρέπει να περάσουμε στην Επιτροπή για τα, <clears throat> για τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπους, που έχει 30 μέρες να αντιδράσει. Μπορούμε λοιπόν να ε, περιμένουμε αυτή την τελική ετοιμιγορία της ΚΡΑΚ μέχρι το Σεπτέμβριο. Για το Διάν, το αντισυλληπτικό αυτό. Έχουμε μια χωριστή διαδικασία που έχει ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου φέτος με αίτηση της Γαλλίας μετά από μια απόφαση να ανασταλεί η εμπορία αυτού του προϊόντος μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Η Γαλλία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια γιατί θεωρεί ότι η σχέση ωφέλους προς το κίνδυνο για την αντιμετώπιση της άκμης ότι είναι αρνητική και θεωρεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες θεραπείες για την ακμή και επίσης έχει εκφράσει ανησυχίες για την χρήση αυτού του φαρμάκου ως αντισυλληπτικού που δεν προβλέπεται για το DIAN. Οι ενδείξεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το προϊόντο αυτό που δεν ε, εγκρίνεται κεντρικά είναι ετερογενής. Για ορισμένα κράτη το χρησιμοποιούν για την καταπολέμηση της ακμής και άλλα κράτη-μέλη ως αντισυλληπτικό. Και επομένως δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα εδώ η διαδικασία είναι πολύ πιο βραχία γιατί είναι νομοθεσία η οποία τέθησε εφαρμογή πέρσι. Μας δίνει μοναχά 60 μέρες για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Εδώ προβλέπουμε λοιπόν το, η Αρμόδια Επιτροπή ΚΡΑΚ να αποφασίσει το Μάιο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσει να περάσει από την Επιτροπή για την Αμοιβαία Αναγνώριση Προϊόντων και επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και την συνεδρίαση της ομάδας ΑΤΚΟ που θα συνεδριάσει 26 Απριλίου. Όσον αφορά τώρα την μνήμα για, ε, για, τα, για η έρευνα που, που χρησιμοποιήθηκε δείχνει ότι το, στον Ταϊάν ε, η χρήση μπορεί να έχει ευρύτερη, ευρύτερη συνέπειες, αλλά είναι ανοιχτή στο κοινό. Όποιος θέλει να συμβάλλει λοιπόν για να εξετάσουμε την αναθεώρηση της χρησιμότητας του ΔΕΑΝ μπορεί να το κάνει. Εμείς απευθυνόμαστε κυρίως σε ασθενείς, υπεύθυνους υγείας και γενικό κοινό. Η συνεισφορά αυτή ε, μπορεί να ληφθεί μέχρι και τώρα. Με αυτά να κλείσω κύρια Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ την, ε, τον φορέα των φαρμάκων. Ευχαριστούμε τον κύριο Βατών και την κυρία Ρέιν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας έχετε παρουσιάσει και πολύ χρήσιμα για τη συζήτησή μας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Κομισιό, στην κυρία Γκιούλουχερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσατε ήδη αρκετά για τις διαδικασίες που εξελίσσονται και την επιστημονική αξιολόγηση που λαμβάνει αυτή τη στιγμή η χώρα ή έγινε στο παρελθόν. Θέλω να επανέλθω στο ρόλο της Επιτροπής στη διαδικασία αυτή. Προφανώς είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η διαδικασία επανεξέτασης όπως και κάθε άλλη τηρεί την νομοθεσία της Ένωσης οτι αυτη η διαδικασια επανεξέταση οπως και καθε αλλη τηρει την νομοθεσια της ενωσης ιδίω, οπως το, το είπε ο κ. Σπετιών την πρόσφατη η νομοθεσία τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Παρακολουθούμε λοιπόν εκ του σύνεγγις ε, την διαδικασία για να την αξιολογήσουμε βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Επίσης, κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ή αξιολογήση, ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ομοιόμορφη νομοθεσία τυχόν μέτρων που προταθούν. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε, να το σημειώσουμε. Οποτεδήποτε ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να έχουμε εναρμονισμένα μέτρα σε όλη την Ένωση. Κάποιοι σημαντικοί παράγοντες ήδη αναφέρθηκαν. Θα επανέλθω σε αυτούς ωστόσο. Είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτό φύση των αδειών των φαρμάκων ε, είναι, όπως γνωρίζετε, είναι διαφοροποιημένη. Τα περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα που εξετάζονται τώρα έχουν τύχη εθνικής άδεια. Λίγα, τρία νομίζω, έχουν κεντρική αδειοδότηση. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί αντικατοπτρίζει κάπως και τη διαδικασία που απαιτείται εκ του νόμου για την αναθεώρηση. Δεύτερο σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πόσο επίγουσα είναι η δράση. Ο κύριος Μετιόν ήδη εξήγησε ότι η μία διαδικασία ακολουθεί αυτή τη στιγμή την ταχύρυθμη τη διαδικασία επίγοντος με μικρό χρονικό διάστημα αναθεώρησης όλων των στοιχείων, κάτι που ξεκινά από την άποψη των γαλλικών αρχών ότι θέλουν σε δύο μήνες να διακόψουν την χρήση του Diane 35 που είναι ένας λόγος διαδικασίας επίγοντος. Η άλλη διαδικασία επιτρέπει περισσότερο χρόνο αναθεώρησης. Ακούσατε τα στοιχεία που αναθεωρηθήκαν ήδη. και εκεί ευτυχώ μπορούμε να κάνουμε μια πιο διεξοδική ανάλυση. Λόγω τη φύση των αδειών και των διαδικασιών πρέπει να ακολουθούν δύο διαφορετικέ οδοί. Εν τέλει δεν έχει σημασία αν ακολουθήσουμε τη διαδικασία του CHMP ή του, της ομάδας συντονισμών, συντονισμού των κρατών μελών. Εν τέλει το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Πρέπει να έχουμε εναρμονισμένη και δεσμευτική νομοθεσία σε ενωσιακό επίπεδο. για να δείξουμε ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση πραγματικά λειτουργεί όπως οφείλει. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν τις επιστημονικές ε, απόψεις και τις κομισιόν και μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Έχουμε διάφορους, διάφορες ομιλήτρες, η κυρία Ροτμπέρεντ, Ζαβόρσκα και πρώτα βέβαια η Λίνα Μακέβαν. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε πρώτα Να ακούσουμε πρώτα τη Φρανσουάς Γκροστέτ, γιατί αυτή ξέρει καλύτερα τι γίνεται στη Γαλλία και θα ήθελα να ξέρω γιατί υπήρξε αυτή η απόσυρση από την αγορά και μπορώ να λάβω το λόγο μετά, αλλά ίσως η Φρονσουάς μπορεί να λάβει το λόγο πρώτη γιατί ξέρει περισσότερα. Φρανσουάς λοιπόν ούτως απεφασίστε, έχει το λόγο. Λοιπόν, θα σας τα πω εντάχει. Υπήρξε μια, ένα μέτρο αναστολής ε, της κυκλοφορίας του Dian 35 στη Γαλλία με, ίσως ε, λόγω του ότι δημιουργήθηκε σάλος καθότι διαπιστώθηκαν κάποια ατυχήματα. Εγώ θέλω να πω, το ξέραμε εδώ και δεκαετίες από την αρχή της ύπαρξης αυτών των ε, ε αντισυλληπτικών που λαμβάνονται με το στόμα, που έχουν κινδύνους. Έχουν κινδύνους. Το να λάβουμε λοιπόν αποφάσεις βάση, ξαφνικά βάσει συναισθηματικών αντιδράσεων είναι επικίνδυνο γιατί στη Γαλλία έχουμε 2,5 εκατομμύρια γυναίκες που, χρησιμοποιούμε, ε, που χρησιμοποιούν ε, ε, αντισυλληπτικά της τέταρτη γενιάς το ίμιση του συνόλου των γυναικών που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά. Δημιουργήθηκε ξαφνικά ένα πανικό στις γυναίκε αυτέ που άρχισαν να λένε να σταματήσω να παίρνω οποιοδήποτε ε, αντισυλληπτικό με όλες τις επιπτώσεις και χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι όχι, μην σταματήσετε μία θεραπεία χωρίς να το ξέρει ο γιατρός. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα πλεονεκτήματα αυτών των ε, αντισυλληπτικών είναι σαφώς περισσότερα από τους κινδύνους που ενέχουν. Μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, όπως ξέρουμε, μπορεί να έχει πολύ πιο δραματικέ συνέπειες για τις γυναίκες. Αυτό είναι το πλαίσιο, να το έχουμε υπόψη μα. Ζητήθηκε λοιπόν από τον Υπουργό Υγείας της Γαλλίας να διακοπεί, να ανασταλεί η κυκλοφορία του φαρμάκου αυτού και προφανώς ε, τέθηκε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιμερισσία Φαρμάκων που χρειάστηκε όπως εξηγήθηκε να, να δώσει μια απάντηση πολύ, σε πολύ βραχή χρονικό διάστημα. Εγώ με κάποιους συναδέλφους πήγαμε στο Λονδίνο και συζητήσαμε για το θέμα αυτό με τους διάφορους ειδικού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Η άποψή μου είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη το αίσθημα πανικού που αναπτύχθηκε χρειάζεται μια ταχύ απάντηση όντως. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεδομένου το ότι ένα αντισυλληπτικό είναι φάρμακο ο συντα... συνταγογράφων εξ και από την αρχή γνωρίζει τους κινδύνους και πρέπει να αξιολογήσει περίπτωση μπροστά σε μια γυναίκα. Αν είναι νέα, αν δεν είναι νέα, που ζητά να χρησιμοποιήσει ένα αντισυλληπτικό, πρέπει να κάνει μια διάγνωση και να διαπιστώσει αν το άτομο αυτό μπορεί να αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κίνδυνο διότι υπάρχει κληρονομικότητα γενετική ή γιατί το άτομο αυτό καπνίζει. Τέλο πάντων, έχει, παρουσιάζει μια σειρά κινδύνων. Ξέρουμε ότι το γεγονός ότι μια γυναίκα καπνίζει είναι αντένδειξη για την χρήση αυτών των αντισυλληπτικών. Το ξέρουν αυτό. Είναι γνωστό. Ας αφήσουμε λοιπόν τις συγκινησιακές αντιδράσεις και ας είμαστε βεβαίως να δώσουμε την πληροφορία και αναφέρθηκε αυτό από τους ε, εκπροσώπους ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Χρειάζεται να παραπέμψουμε στην ε, νομοθεσία. Έχουμε τα κείμενα της φαρμακοεπαγρύπνησης, ας τα εφαρμόσουμε, αλλά ας ελέγξουμε την πληροφορία. Ο ρόλος του συνταγογραφούντος είναι πολύ σημαντικός. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε σαφή, γρήγορη απάντηση, διότι πρέπει να πάψει αυτό το αίσθημα ασφάλεια που αισθάνονται πολλές γυναίκες. Στη Γαλλία σίγουρα, ίσως και αλλού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, κατά πόσον πρέπει η ασυνταγογράφηση να ακολουθεί την ε, διαπίστωση των κινδύνων για αυτά τα δεύτερα, φάρμακα δεύτερη, τρίτης, τέταρτη γενιάς είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Κατά την άποψή μου, η απόφαση των γαλλικών αρχών να, να αναστείλουν την κυκλοφορία είναι λάθος, αλλά πρέπει να το πούμε σαφώς. Διότι χρειάζεται να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Είναι σημαντικό για όλες τις γυναίκες που χρησιμοποιούν αυτό το είδος αντισύλληψης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ η Λίντα. Ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να ξέρω ποια είναι η κατάσταση στη Γαλλία, γιατί οι δικές μου πληροφορίες ήταν λιγάκι μπαγιάτικες πριν από μερικές εβδομάδες. Βλέπω ότι μονάχα ένας άνδρας βουλευτής είναι παρόν εδώ. Είναι ενδιαφέρον ότι η σύλληψη είναι ένα γυναικείο πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε εμείς μεταξύ μας. Ναι, κοιτάξτε. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Βέιν Ρέιν να μας πει το εξή και να το πει δημοσίως, γιατί μας δώσατε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά αντισυλληπτικών και μας είπατε ότι η τρίτη και η τέταρτη γενιά επέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τη δεύτερη γενιά για το πρόβλημα αυτό της τρόμβωσης. Φυσικά όλα αυτά είναι γνωστά. Γιατί έχουμε τότε τρίτη και τέταρτης γενιάς. Γιατί πάρα πολλέ γυναίκε θα πούν αν είναι μεγαλύτερο ο κίνδυνος. Γιατί να τα χρησιμοποιήσουν. Είναι καλύτερα αυτά τα αντισυλληπτικά από άλλε πτυχές από τα αντισυλληπτικά δεύτερη γενιάς. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσει κανείς όταν πηγαίνει να ζητήσει αντισυλληπτικά από τον γιατρό. Γιατί λοιπόν τα αντισυλληπτικά τρίτη και τέταρτη γενιά είναι καλύτερα, γιατί τα αφήνουμε να κυκλοφορούν στην αγορά εάν αυτά της δεύτερης γενιάς για αυτό το θέμα είναι καλύτερα. Μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για άλλα θέματα. Το δεύτερο θέμα είναι όλη αυτή η αντιμετώπιση των αποκεντρωμένων, της αποκέντρωσης για την παραγωγή των προϊόντων και την εμπορία τους. Και στη Γαλλία υπήρχε και πρόβλημα ότι χρησιμοποιούταν το DIAN ε, ως αντισυλληπτικό αντίθετα από αυτό που έλεγε η ετικέτα του. Εγώ θα ήθελα να ξέρω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε για αυτά τα θέματα. Οι καταναλωτές στην Ευρώπη περισσότεροι εντυπωσιάζονται και σοκάρονται όταν οι οδηγίες χρήσης λένε διαφορετικά πράγματα στη Γαλλία από ό,τι στην Αγγλία. Ναι, το ίδιο φάρμακο θα πρέπει να έχει λογικά την ίδια πληροφορία. Και ξέρω ότι έχω αναφέρει το πρόβλημα αυτό και στο παρελθόν για τα φαρμακευτικά συσκευάσματα τα παιδιά που κάποια επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, κάποια δεν χρησιμοποιούνται. Και όταν ταξιδεύουν από τη μια χώρα στην άλλη οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πώς, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Όταν ανακύπτουν τέτοια προβλήματα. Και το τελευταίο μου ερώτημα. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν ε, αναφέρει προβλήματα, νέα προβλήματα για τα ε, αντισυλληπτικά που λαμβάνονται ε, από το στόμα. Γνωρίζετε να υπάρχουν άλλες ε, χώρες που είχαν απρόπτα ε, συμπτώματα από τη χρήση αυτών των ε, αντισυλληπτικών. Ελπίζω ότι καταγράφετε όλα αυτά τα ερωτήματα. Η Μισελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μετά από αυτά που ρωτάει η Λίντα, εγώ θα σας δώσω συγκεκριμένα δεδομένα από τη Γαλλία. Πρώτον, το σκάνδαλο αυτό ξεκίνησε μετά από μια προσφυγή. Η Μαριόν Λαρά υπέβαλε προσφυγή διότι είχε πρόβλημα θρόμβωσης. Και μετά επειδή είχε χρησιμοποιήσει τέταρτη γενιά αντισυλληπτικό. Μετά από αυτή την περίπτωση είχαμε 700 προσφυγές από διάφορες Γαλλίδες οι οποίες είχαν τέτοια προβλήματα εμβολή. Σήμερα, σήμερα το πρωί ακόμα, η Γαλλική Υπηρεσία Φαρμάκων ε, παρουσίασε μία μελέτη για όλα τα αντισυλληπτικά. Πρόκειται για 4.700.000 και διαπίστωσε ότι υπήρχαν 2.000 και ατυχήματα θρόμβωσης στο αίμα, 20 πρώιμοι θάνατοι, 14 από τους οποίους οφείλονται σε αντισυλληπτικά τρίτης και τέταρτης γενιάς. Σήμερα το πρωί, φρέσκια μελέτη. Τι δείχνει, δείχνει ότι από το 2000 μέχρι το 2011 είχαμε 20 περίπου θανάτους, εκ των οποίων 14 οφείλονται στα αντισυλληπτικά αυτά τρίτης και τέταρτης γενιάς. Αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί είναι ότι χρειάστηκε μια προσφυγή για να τεθεί το ζήτημα αντισληπτικών τρίτης και τέταρτης γενιάς. Ενώ αν κοιτάξουμε τι γίνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε. Σήμερα στι Ηνωμένε Πολιτείε έχετε 13.500 προσφυγέ οι οποίε έχουν κατατεθεί για την χρήση αντισληπτικών τρίτη και τέταρτη γενιά. Το 2011 στην Ελβετία ήδη είχαν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες αρχές σχετικά με το θέμα γιατί δίνουμε σε νέες γυναίκες τέτοια της λεπτικά τρίτης και τέταρτης γενιάς που δεν έχουν πρόβλημα ε, με κάπνισμα ούτε κανέναν άλλον κίνδυνο έχουν όμως τελικά προβλήματα ε, θρόμβωσης. Η Λίντα λέει γιατί δεν υπάρχουν περισσότεροι άντρες εδώ. Ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που παίρνουν τα αντισυλληπτικά αυτά και το πρώτο θέμα που τίθεται είναι πώς είναι δυνατόν. Και αυτό θέλω να ρωτήσω στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Στις Ηνωμένε Πολιτείες σας είπα 13.500 προσφυγές. Στην Ελβετία, σε άλλες χώρες. Παρόλα αυτά δεν έγινε νέα αξιολόγηση κινδύνων για τα αντισληπτικά τρίτης και τέταρτης γενιάς στην Ευρώπη. Έπειτα, υπάρχει το θέμα του φαρμάκου Dian 35. Το Dian 35 τι έχει, έχει την άδεια για να κυκλοφορεί για φάρμακο, ως φάρμακο κατά της ακμής, όχι όμως ως αντισυλληπτικό. Ιανουαρίου 2013 113 περιπτώσεις θρομβώσης από τα γενώσιμα φάρμακα μετά τον Διάν. Άρα υπάρχει καταγραφή του προβλήματος. Γιατί όμως πρέπει να γίνει προσφυγή τελικά για να τεθεί το ζήτημα του Διάν 35. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει πρόβλημα για να σκεφτούμε, α, μήπως υπάρχουν παρενέργειες. Και τώρα όταν μια νέα γυναίκα πάει σε ένα γιατρό, σε ένα γυναικολόγο και δεν πρέπει να σκεφτούμε πρώτα να της δώσουμε δεύτερης γενιάς αντισληπτικό πριν σκεφτούμε τα τρίτης και τέταρτης. Εγώ έχω πρόβλημα με την φαρμακοεπαγρύπνηση, γιατί διαπιστώνουμε ότι όταν οι νέες αυτές γυναίκες πρέπει να σκεφτούν, έτσι, μήπως το πρόβλημα το που είχαν έχει να κάνει με το χάπι που πήρανε. Αυτό δεν πρέπει να το σκεφτούν τις παρενέργειες, δηλαδή οι επιτροπές φαρμακοαπαχρύπνησης. Τελικά οι ασθενείς δεν ενημερώνονται για το ότι μπορούν να απευθυνθούν στη φαρμακοπαχρύπνηση. Τα, τις παρενέργειες δηλαδή δεν τις μαθαίνουμε αρκετά. Πώς θα βελτιωθεί λοιπόν αυτή η φαρμακοπαχρύπνηση και πώς θα κάνουμε τους γιατρούς να ενημερώνουν για τις παρενέργειες όπω και στο προηγούμενο σκάνδαλο, οι χειρούργοι ήταν εκείνοι οι οποίοι τελικά το έθεσαν, αλλά μετά από καιρό. Αν γίνεται έγκαιρα, θα αποφεύγονται καθυστερήσει και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε που έχουν πάρει τα αντισληπτικά τρίτη και τέταρτη γενιά. Και επανέρχομαι στο Dian 35. χώρε όπω οι κάτω χώρε επιτρέπουν το Dian 35 ω αντισληπτικό. Στη Γαλλία χρησιμοποιόταν όπω και με το Mediator. Χρησιμοποιόταν μόνο για την ακμή είτε το DIAM 35 είναι προβληματικό ακόμα και για την ακμή, οπότε το απαγορεύουμε, ή θα πρέπει να πούμε χρησιμοποιήστε το για την ακμή, αλλά για μικρά χρονικά διαστήματα, γιατί μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να συλλάβετε παιδί. Υπάρχουν χώρες δηλαδή που το χρησιμοποιούν και για την ακμή και ως αντισληπτικό, άλλες που το χρησιμοποιούν μόνο για την ακμή, αλλά καμιά φορά και για την ακμή, χωρίς όμως να έχει πάρει άδεια στις χώρες αυτές για αντισυλληπτικό. Συνεπώς, επιτρέψτε μου να το πω, πρέπει σε όλες τις χώρες να ρωτήσετε τι χρησιμοποιούν οι γιατροί. Οι επαγγελματίες, οι γιατροί πρέπει να φροντίσουν πρώτα να δίνω την ενημέρωση για τις παρενέργειες. Εκεί υπάρχει η πρώτη αδυναμία. Και έπειτα φυσικά και πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση για τα αντισυλληπτικά τρίτης και τέταρτης γενιάς. Γιατί σας τα έδωσα τα νούμερα παρά αυτά που λέει η κυρία Γκροστέτ. Έχουμε δυο φορές παραπάνω προβλήματα από τα αντισυλληπτικά τρίτης και τέταρτης γενιάς από ότι για εκείνα δεύτερης γενιάς. Άρα υπάρχει πρόβλημα ουσία εδώ. Ευχαριστώ, Μισε. Η Άννα Ρόσπα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω, θα είμαι σύντομη, αλλά να πω καταρχάς ότι συμφωνώ με τη Λίντα. Ε, μόνο γυναίκες είναι εδώ, αλλά τα, χά, τα χάπια αυτά τα παίρνουμε λόγω των ανδρών. Μην το ξεχνάμε. Να σας πω ξεκάθαρα, η ζωή είναι επικίνδυνη. Είτε παίρνεις το χάπι είτε δεν το παίρνεις. Το αντισυλληπτικό χάπι ωστόσο έχει αλλάξει επαναστατικά την κοινωνία τα προηγούμενα 60 χρόνια. Οι γυναίκες για πρώτη φορά ε, μπορούν να αποφασίσουν για τη ζωή τους. Αυτό έγινε αφού άρχισαν να διατίθενται αυτά τα αντισυλληπτικά χάπια. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να καταλάβουμε καλά την κατάσταση. Ε, όταν ε, μίλησα με τις ε, δανεικές αρμόδιες αρχές, την ε, εντύπωση ότι το χειρότερο είναι το χάπι τρίτης γενιάς. Άρα χρειάζεται να εξεταστεί το θέμα και να διδαχθούν οι γιατροί μας ότι πρέπει να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για τους παράγοντες κινδύνου. Βεβαίως, πρόκειται για ορμονικές παρασκευές. Αλλά δεν είναι αυτό που εν τέλει ε, καταπίνουν οι γυναίκες. Η ερώτηση που έχω λοιπόν είναι υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σαφή που συγκρίνουν την αύξηση του κινδύνου καρκίνου ή εμβολής για γυναίκες όταν χρησιμοποιούν άλλα φάρμακα, αντικαταθλιπτικά για παράδειγμα, ή ενέσιμα ναρκωτικά, ή νόπνευμα. οδηγούν αυτά σε αύξηση του κινδύνου. Και μιλάμε για καπνιστές, αλλά και άλλα στοιχεία αποτελούν, που αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας, που επηρεάζουν το πώς αντιδρούν τα φάρμακα. Υπάρχουν λοιπόν συγκριτικές στατιστικές. Ευχαριστώ. Η ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι σίγουρη τι κάνουμε ακριβώς εδώ θα χαιρόμουν αν καταλαβαίναμε όλοι ότι είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την εντύπωση ότι εστιάζουμε μονάχα σε ένα γαλλικό πρόβλημα. Εγώ έχω βαρεθεί να αντιμετωπίζω αυτό το θέμα. Αντιμετωπίστε τα προβλήματά σας όταν θεωρείτε ότι μπορείτε να δίνετε εθνικέ εγκρίσει. Αυτό θα έλεγα στου Γάλλους. Αν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό εθνικά, τότε μπορώ να καταλάβω. Γιατί πιστεύω σε μια κεντρική διαδικασία έγκριση. Αλλά η διαδικασία, όπω αναφέρθηκε από του εκπροσώπους τη ΕΜΑ, είναι μια βαριά διαδικασία που ξέρουμε ήδη α, εδώ και 30 χρόνια από όλε τι γενιέ των συνδυασμένων αντιληπτικών, το ξέραμε όλοι μας Σχεδόν όλες οι γυναίκες αυτή την αίθουσα έχουν χρησιμοποιήσει αντισυλληπτικά σε κάποια φάση της ζωής τους. Ξέραμε όλοι ότι υπήρχε ο κίνδυνος θρόμβασης. Το ξέραμε όλες. Και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε την ευθύνη αλλού από τους γυναικολόγους. Μπορεί να πει κανείς δεν τα εγκρίνει αυτά τα αντισυλληπτικά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω ποιος θα συμφωνούσε με μια τέτοια αρρύθμιση. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν διάφορες μορφές αντισυλληπτικών όλες μας και θα ήθελα να υπάρξει μια πραγματική έρευνα για τα θέματα αυτή. Όλα τα φαρμακευτικά ε, προϊόντα έχουν παρενέργειες. Εγώ πήρα για έξι χρόνια βαριά φάρμακα που έπρεπε να τα πάρω και είχε τεράστια, τεράστιες παρενέργειες. Αλλά η επιλογή μου ήταν να τα πάρω αυτά και να ελπίσω ότι θα επιβιώσω ή να μην τα πάρω και να μειώσω τις δυνατότητες επιβίωσης. Πάντα έχουμε λοιπόν μια ισορροπία. Ίσως θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο ουδέτεροι. Μιλάμε για διαφορετικές διαδικασίες, κεντρική διαδικασία έγκρισης και εθνική διαδικασία έγκρισης για τα φάρμακα. Εγώ νιωθώ πολύ άνετα γιατί είμαι εναντίον των εθνικών συστημάτων έγκρισης. Πίστευα ότι μόνο πρέπει να υπάρχει μια κεντρική διαδικασία έγκρισης. Φυσικά η αίμα θα είχε όλη την ευθύνη τότε ο Οργανισμός Φαρμάκων του Λονδίνου. Προς το παρόν όμως δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές να γίνει εθνική έγκριση. Έχουμε το ίδιο ενεργό συστατικό το οποίο χρησιμοποιείται σε ένα κράτος μέλος για να, αντιμετωπίζονται, ε, να αντιμετωπίζεται η ακμή και σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται αυτό το ειδικό, αυτή η ενεργή ουσία για αντισυλληπτικό που λαμβάνεται από το στόμα. Αυτό είναι μέσα στη δυνατότητα των εθνικών αρχών να το κάνουν αυτό. Μα αυτό είναι τρέλα, καθαρή τρέλα. Και αν πούμε ότι δεν πρέπει να εγκρίνεται για την αντιμετώπιση της ακμής αλλά μόνο σαν αντισυλληπτικό, μα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μέσα στα 540 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναικολόγοι και οι δερματολόγοι θα σεβαστούν αυτήν την εντολή. Υπάρχει πάρα πολλές φορές ε, ε, η χρήση προϊόντων αντίθετα από τις οδηγές χρήσης από τους ε, δερματολόγους. Γιατί τους λένε έχω αυτό το αντισυλληπτικό το οποίο όμως δουλεύει μούρλια για την ακμή. Θέλετε να το πάρετε ή όχι. Αυτή η χρήση λοιπόν των φαρμακευτικών προϊόντων δεν μπορεί να αποφευθεί τελείως. Δεν μπορούμε να πούμε σε κάθε ιατρείο και σε κάθε κλινική και να τους ελέγχουμε τους γιατρούς. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς τα φάρμακα από αυτούς που προβλεπόταν. Και οι παιδίατροι το κάνουν αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν υπήρχαν ειδικά παιδιατρικά φάρμακα. Το δέχονται και σε επίπεδο δεοντολογίας οι γιατροί. Αν είσαι 20 χρονών, δεν έχει τον ίδιο με μια 40, επομένω σου δίνουμε αυτό το φάρμακο. Επομένως, Τίποτα από όλα αυτά που συζητούμε είναι καινούριο. Γιατί η Γαλλία αποφάσισε να αντιδράσει, η Φρανσουάζ το είπε αυτό ότι είναι κάτι συγκινησιακό, εγώ νομίζω ότι είναι μια ενέργεια τύπου ποντίου πιλάτου απέκτησης της ευθύνης. Μα η Γαλλία έχει την ευθύνη αυτή. Τέρμα. Και το θέμα είναι, θέλετε να κατανοήσετε ότι τα αντισυλληπτικά τέταρτη γενιάς, τα οποία είναι τα μόνα που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ορισμένη κατηγορία γυναικών, ότι δεν θα είναι διαθέσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Όσο δεν έχουμε λοιπόν μια σαφή διαδικασία, είναι καλύτερα να είναι κεντρική, τουλάχιστον να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά εμεί δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τι εθνικέ αρχέ να πάνε προ αυτή την κατεύθυνση δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τη Γαλλία και τη Γερμανία να έχουν τα ίδια, τις ίδιες οδηγίες χρήσεως, γιατί ξεφεύγουμε από τις αρμοδιότητές μας. Και όσο δεν το κάνουμε αυτό, οι γυναικολόγοι και σε αυτήν την περίπτωση και οι δερματολόγοι δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα φάρμακα. Και η φαρμακοεπαγρύπνηση δεν προβλέπεται για τέτοιου είδους διαδικασίες. Ξέρουμε ήδη ότι υπάρχουν θρομβώσεις ως παρενέργειες των αντισυλληπτικών. Δεν έχει δημιουργηθεί η διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης για αυτά τα θέματα, αλλά μόνο για άγνωστες παρενέργειες. Μα υπάρχουν ήδη και στις οδηγίες χρήσεως. Αν έχει κανείς μεγάλο βάρος, αν καπνίζει κανείς πολύ, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Το ξέρουν όλοι. Τελικά λοιπόν, όσο έχουμε ακόμα εθνικά συστήματα έγκρισης και όταν έχουμε διαφορετικούς εθνικούς φορείς που έχουν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα και πολύ διαφορετική ποιότητα. Και όσο επιτρέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν εθνικές διαδικασίες έγκρισης με διαφορετική έγκριση για διαφορετική διάγνωση και ξέρουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς τα φάρμακα, τέτοια προβλήματα θα παραμείνουν. Μόνο δύο συμβουλές μπορώ να σας δώσω ή να καταργήσετε τις εθνικές διαδικασίες έγκρισης και αυτή είναι η δική μου πρόταση. Ή απλώς να δεχτούμε ποια είναι η κατάσταση. Αλλά δεν θέλω οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης να μας δημιουργούν προβλήματα γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει ο Εθνικός Φορέας ή αλλιώς να το καταργήσουμε και να τελειώνει πια. Ευχαριστώ την κυρία Ροτ Μπέρεντ. Η Εστέρ Ντελάγκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, όπως είπε και η Λίντα Μακέβεν, κοιτάξτε την αίθουσα. Πράγματι, αυτή τη στιγμή που συζητάμε για θέματα αντισυλληπτικών, μόνο γυναίκες έχουν μείνει στην αίθουσα. Εγώ έστειλα και με το Twitter και όντως γυναίκες αντιδρούν. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Στην Ολλανδία πράγματι μισό εκατομμύριο γυναίκες παίρνουν αντισυλληπτικά. Είναι αναμενόμενο. Άκουσα τι είπε η Dagmar Μπέρεντ για τις διάφορες διαδικασίες. Ναι, αλλά τελικά ποιο είναι το μήνυμα. Το τι συμβαίνει στη Γαλλία ήταν γνωστά πράγματι τα δεδομένα και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και είναι η ηλικία ακριβώς που ασχολούμαστε κι εμείς με τα θέματα αυτά και στις ειδήσει. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι τα δυσλειπικά τρίτης, τέταρτης γενιάς ε, λοχεύουν κινδύνους για θρόμβωση, ε, αλλά έχουν λιγότερους κινδύνους όσον αφορά την δημιουργία καρκίνων. Οπότε πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας ε, και τα δύο. Το θέμα της εθνικής ε, διαδικασίας έγκρισης ή της κεντρικής, της ευρωπαϊκής είναι κάτι όμως που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ γιατί καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στον κόσμο που το ακούει. Είναι μεγάλη η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Οι συζητήσεις που γίνονται εδώ είναι πολλαπλές. Είναι το θέμα της έρευνας, είναι το θέμα της συνταγογράφησης και είναι και το θέμα της εμπορίας. Και πώς δηλαδή σε καθημερινή βάση χρησιμοποιεί τα φάρμακα αυτά η κάθε γυναίκα. Όσον αφορά την έρευνα, εδώ είναι πολύ βασικό να γίνεται η έρευνα για την θρόμβωση. Χρηματοδοτείται όμως από τη φαρκοβιομηχανία και σε μερικές περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν ότι δεν αυξάνει ιδιαίτερο κίνδυνος για θρόμβωση. Από ανεξάρτητες όμως έρευνες έχουμε αποτέλεσμα ότι πρόκειται για διπλασιασμό των θρομβώσεων. Οπότε τελικά ε, πρέπει να ξέρουμε και ποιος κάνει τις έρευνες κάθε φορά για να καταλήξουμε σε, μια, σε ένα ισορροπημένο συμπέρασμα. Τι απ' όλα ισχύει δηλαδή όταν κανείς παίρνει τα αντισυλληπτικά αυτά τρίτη και τέταρτη γενιά και να τα συγκρίνουμε με τα αποτέλεσματα των ερευνών από τη δεύτερη γενιά. Η συνταγογράφηση τώρα είπαμε ότι οι γυναικολόγοι συνταγογραφούν. Στην Ολλανδία όχι, είναι ο πρακτικό γιατρός, ο παθολόγος, ο γενικό γιατρός όπως τον λέμε εμείς που βασίζεται στην πιεσή σας, κάνει κάποιες βέβαια εξετάσεις από τα 17, 18 και 16 ακόμα μια Ολλανδέζα αρχίζει να έχει σεξουαλική ζωή. Μπορεί λοιπόν πάρα πολλά χρόνια να το παίρνει, μέχρι τα 38 για παράδειγμα. Μπορεί να παίρνει τέτοια δυσλεπτικά χωρίς να έχει πάει ποτέ σε γυναικολόγο μια γυναίκα στην Ολλανδία, ε? μόνο στον γενικό της παθολόγο. Έτσι γίνεται. Και βλέπω ότι με κοιτάτε με ανοιχτά τα μάτια και όμως έτσι είναι. Μόνο ο γενικός σας παθολόγος μπορεί να σας συνταγογραφήσει τα αντισυλληπτικά στην Ολλανδία. Δεν χρειάζεται να πάτε σε γυναικολόγο. Αν ξέρω στο Βέλγιο είναι αλλιώς. Πάντα ε, πρέπει να πάτε σε γυναικολόγο. Είναι διαφορετική ίσως και η κατάρτιση, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετική ενημέρωση που παίρνει κανείς από τον παθολόγο του και διαφορετική αυτή που παίρνει από τον γυναικολόγο του. Στην Ολλανδία έχει γίνει μία μελέτη για την ε, χρήση ε, προϊόντων και εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε για τα αποτελέσματα μελετών που έχουν γίνει σε σχέση με τα τηλεπτικά δεύτερης και τρίτης γενιάς, κατά πόσο τα αποτελέσματα αυτά τελικά δείχνουν πραγματικά ε, συμπεράσματα ή ε, είναι πρόκειται για χειραγώγηση που έχει γίνει όσον αφορά. Γιατί βλέπουμε ότι αλλού έχουμε έρευνες που καταλήγουν στο συμπέρασμα για διπλασιασμό των ε, κινδύνων θρόμβωσης και αλλού όχι. Στην Ολλανδία λοιπόν θα έπρεπε κανονικά να έχουμε καταλήξει στην προτίμηση των συντεσλεπτικών δεύτερης γενιάς. Έχουμε μιλήσει και εμείς κατά του Dian 35, αλλά όχι για τα αντισλεπτικά τρίτης και τέταρτης γενιάς. Παρ' όλα αυτά, το 1 τρίτο των ε, γυναικών στην Ολλανδία χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά τρίτη και τέταρτη γενιά. Ενώ θα έπρεπε να ξέρουν οι γενικοί παθολόγοι ότι δεν πρέπει να δίνουν προτίμηση στα αντισυλληπτικά τρίτη και τέταρτη γενιά. Δεν συμβαίνει όμω αυτό, ή τουλάχιστον στην πράξη δεν ισχύει. Θα έπρεπε να υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες για τη συνταγογράφηση τέτοιων αντισυλληπτικών όχι μόνο να είναι γνωστά τα αποτελέσματα των μελετών, αλλά να υπάρχουν κατευθυντήριε γραμμέ για τη συνταχογράφηση. Αυτά ήταν για το δεύτερο σκέλο τη συνταχογράφηση. Και έρχομαι στο τρίτο επίπεδο τη συζήτηση, που πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα, αυτό είναι το θέμα τη εμπορία. Μιλήστε με τι γυναίκε γιατί παίρνουν το, 30, το Dian 35 ή το Γιασμίν, που είναι τέταρτη γενιά πολύ σε ονομασίες έτσι, έτσι όπως λέγονται, ενώ άλλα αντισληπτικά δεύτερης γενιάς έχουν κάτι πολύ επιστημονικά ονόματα, τι θα πούνε, θα πούνε γιατί είναι πιο ελαφρύ αντισυλληπτικό αυτό. Και όλοι λένε ότι βοηθούν στην ακμή και δεν χοντρένουν, δεν σαπαχαίνουν. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ο παραγό του Γιασμίν κάνει αυτή τη διαφήμιση και ένα 1,2 δις όμως έχουν πληρωθεί σε αποζημιώσεις επειδή πολλές γυναίκες έχουν παρασυρθεί από τη διαφήμιση αυτή ενώ επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο ότι δεν σε παχαίνει. Άρα είναι θέμα διαφήμισης. Πώς ε, πάει στην εμπορία ότι δεν έχει άνδρο, ορμόνες τέτοιες ε, πολλές. ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά ως προς αυτό με τα αντισλεπτικά δεύτερης γενιάς. Άρα είναι το πώς το πουλάς το προϊόν. Είναι πολύ ενδιαφέρον για τις γυναίκες να ακούνε ότι δεν θα παχύνουν. Αυτό μένει πιο πολύ στο μυαλό τους παρά ο κίνδυνος για θρόμβωση. Ακόμα και για αυτούς που παίρνουν πολύ συχνά το αεροπλάνο, κανονικά πρέπει να υπάρχει αντίδειξη. Οπότε, ακόμα και στο iPad, καθημερινά αυτό κοιτάει ο κόσμος. Αν κοιτάξει για αντισυλληπτικά στην Ολλανδία, φτάνει σε ένα site που λέγεται αντισυλληπτικά NL. Είναι όμως κάτι το οποίο χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία για μας αυτό είναι κάποιο είδους διαφήμιση που θα έπρεπε να απαγορεύεται. Όμως η επιθεώρηση στην Ολλανδία είπε ότι δεν πρόκειται για διαφήμιση, αλλά πρόκειται για ενημέρωση που δίνεται ελεύθερα. Ε, διαβάστε τι λέει για το Γιασμίν. Λέει ότι είναι ένα ε, πιο ελαφρύ αντισυλληπτικό που βοηθά στο να μην παχαίνεις. Με εκεί το πρόβλημα. Γιατί αυτό εξηγεί στο κάτω-κάτω γιατί οι γυναίκες εξακολουθούν και πηγαίνουν στον ε, παθολόγο τους και ζητάνε συνταχογράφηση για τα αντισυλληπτικά τους. Τελικά ζητούν να τους γράψουν ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να ελοχεύει μεγαλύτερο κίνδυνο για μία πτυχή αλλά όχι για άλλε. Λοιπόν, συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο πολύ, αλλά πιστεύω ότι εδώ πέρα όντω έχουμε τρία επίπεδα και θα έπρεπε να αναλυφθεί δράση και στα τρία αυτά επίπεδα από του διάφορου αρμόδιου. Ευχαριστώ. Ναι, ήταν πράγματι μακροσκελής η Άννα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω ήδη αναφέρθηκαν. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν ότι οι ανεπιθύμητες παρενέργειες των αντισυλληπτικών είναι γνωστά εδώ και πολλή χρόνια. Ίσως δεν τα προσέξαμε επαρκώς ξεκινήσαμε να δούμε όταν διαπιστώσαμε μια πολύ δραματική κατάσταση. Επιπτέον, επιπλέον, όταν οι αλλαγές ήταν, οι επιπλοκές ήταν τόσο σύνθετες που δεν μπορούσες να τις αγνοήσεις, διότι εν τέλει οδηγούσαν στο θάνατο, δεν μπορούμε να γνωρούμε το ότι υπάρχουν παρενέργειες που δεν τις διαπιστώνει ο, ασθενή, ο ιατρός ή ο ασθενής. Μπορεί ο ασθενής ε, να είναι μια νέα κοπέλα που να θέλει απλά τη σύλληψη και ο γιατρός να μην σκέφτεται ότι τόσο νέο άτομο μπορεί να πάθει εγκεφαλικό. Ε, κάτι άλλο οι ανεπιθυμίτες παρενέργειες είναι πιο συχνές στις γυναίκες που έχουν μια γενετική προδιάθεση, ας πούμε για προδιάθεση δημιουργίας θρομβικών επεισοδίων. Μια νέα γυναίκα κανονικά που ξεκινά να παίρνει το χάπι. Θα ρωτήσει από πριν το γιατρό της. Ίσως αυτός να είναι γυναικολόγος. Συνήθως εκεί γίνεται η πρώτη επαφή στις περισσότερες χώρες. Κατόπιν ο γυναικολόγος θα εξετάσει όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κοπέλα. Θέλω να υπογραμμίσω ωστόσο ότι αυτό είναι το ιδεώδες. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου η αντιβίωση ή η, αντι, συγγνώμη, η αντισύλληψη μπορεί να δίνεται με, οποιαδήποτε, με συνταγογράφηση από οποιοδήποτε ε, γιατρό και συχνά βρίσκει κανείς ε, παραπλανητικές πληροφορίες στο ίντερνετ και οι γυναίκες αποφασίζουν να πάρουν το α ή β αντισυλληπτικό βασιζόμενες σε αυτές τις πληροφορίες. Κάτι δε που είναι ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι συχνά οι γιατροί δεν το αντιμετωπίζουν επαρκώς σοβαρά, ούτε αναφέρουν τις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Πιστεύω λοιπόν ότι μία ευρωπαϊκή ρύθμιση που δεν χρειάζεται να είναι λεπτομεριακή αλλά πρέπει να καλύπτει τα βασικά θέματα είναι ευκταία. Σε μια τέτοια περίπτωση τα αντισυλληπτικά θα μπορούσαν να συνταγογράφονται πάντα από γιατρό. Η απόφαση για το κατά πόσον αυτό το αντισυλληπτικό είναι το ενδεδειγμένο ή όχι για τη γυναίκα πρέπει να είναι απόφαση του γυναικολόγου. Ένα, μάλλον είναι γεγονός ότι αυτά τα αντισυλληπτικά έχουν προβλήματα για γυναίκες που έχουν προδιάθεση και ότι θα πρέπει να γίνονται γυναικολογικές εξετάσεις προγενέστερα. Επίσης θα πρέπει να γίνονται και κάποιες γεννητικές εξετάσεις για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη μεγαλύτερη ευαισθησία. Το άλλο θέμα που μπορούμε να δούμε είναι η πολιτική επιρροή των φαρμακευτικών ε, εταιριών. Και βέβαια το ερώτημα είναι, δεν, το, δεν είναι δήλωση αυτό που λέω, ερώτημα είναι, η πολιτική πολιτική απόφαση σε ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο χρειάζεται. Το Κοινοβούλιο πρόσφατα υιοθέτησε ένα κείμενο για ε, ενδοκρινολογικούς ε, διαταρακτές, διαταράκτες που έχουν επιπτώσεις ε, στην ορμονική αντισύλληψη. Πιστεύω ότι η Ένωση θα πρέπει να κάνει μια παντίστοιχη έκθεση όπως αυτή της της έκθεσης που κάνει η Σουηδία για τα για τις, αντε, για τις, παρενέργειες, τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των αντισυλληπτικών. Ε, Είτε από την άποψη της τοξικότητας ή από την άποψη της ε, διατήρησης της ε, συνέχιση της παρουσίας των ε, διαταρακτών αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέγει πρόεδρος. Κύριε Κοντέτ και η κυρία Ριβάλτη θέλουν να επανέλθουν. Κροστέτ και Ριβάλτη. Αλλά πάρα πολύ σύντομα για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Ένα λεπτό μονάχα, η καθεμία σας. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν ε, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για σκάνδαλο, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με σκάνδαλο. Δεν επιτρέπω να το λέμε αυτό. Υπάρχει μια προσφυγή στη Γαλλία και μετά από την προσφυγή αυτή, μια υπουργό που πανικοβλήθηκε, αμέσως ζήτησε πληροφορίες και στο μεταξύ ε, απαγόρευσε την κυκλοφορία προσωρικά. Πιστεύω ότι δεν έπαιξε το ρόλο που έπρεπε να παίξει. Εγώ συμφωνώ με την Dagmar Ροτμπέρετ για το ότι θα έπρεπε να περάσουμε σε έναν κεντρικό οργανισμό φαρμάκων όπου όλες οι γυναίκες ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκονται επίσης ώρες. Πιο συγκεκριμένα για το 35 έχει άδεια για αντιμετώπιση της ακμής. Άρα δίνεται για σύντομα χρονικά διαστήματα. Δεν συνταγογραφεί κανείς για χρόνια τη θεραπεία της ακμής. Εντάξει, μου κάνω νόημα ότι πρέπει να σταματήσω, αλλά να ξέρουμε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Μην μιλάμε για σκάνδαλο, γιατί πάντα γνωρίζαμε από την αρχή ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Ήταν γνωστό αυτό. Και τώρα ζητάμε από τους επαγγελματίες της υγείας, από αυτούς που γράφουν, να αναλάβουν την ευθύνη. Ναι, να το κάνουν. Αυτό πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Κύριε Μίσελ, θέλω να απαντήσω κι εγώ σε πολλές ε, παρεμβάσεις. Δεν είναι γαλλο, γαλλο, γαλλικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, γιατί μιλάμε για τα αντισυλληπτικά τρίτη και τέταρτη γενιά. Αυτό δεν είναι καθαρά γαλλικό θέμα. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και φάνηκε ότι υπάρχει έλλειψη πληροφορίας. Δεύτερον, ότι οι γιατροί, οι γυναικολόγοι, οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι στα νέα φάρμακα, αυτοί είναι που δίνουν τα φάρμακα τρίτης και τέταρτης γενιάς γιατί είναι τα πιο πρόσφατα και θεωρούσαν τα λιγότερα προβληματικά. Τώρα αρχίζουν να ανακρούν πρίπνα. Το θέμα δεν είναι η κεντρική ή η εθνική έγκριση και επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Το θέμα είναι η νέα αξιολόγηση κινδύνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει οι πληροφορίες να έρχονται από τα φαρμακευτικά εργαστήρια, γιατί είναι και δικαστές και διάδικοι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και θα πρέπει να εμπλέξουμε περισσότερο και να συνειδητοποιήσουμε τους ε, ιατρούς και τους ε, ασθενείς, ώστε τα θέματα αυτά να μην έρχονται μόνο από τα φαρμακευτικά εργοστάσια. Κύριε Παρβάνοβα, σύντομα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό είναι μερικές φορές να είσαι τελευταίος. Και εγώ σκεφτόμουν τι κάνουμε εδώ σήμερα και γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση. Τι δυνατότητες έχουμε εμείς ως νομοθέτες να επέμβουμε στο ζήτημα αυτό. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το ένα προκύπτει από τη μαζική χρήση αντισυλληπτικών. Το άλλο από την έλλειψη σωστών ιατρικών πρακτικών που είναι συμβατές σε όλα τα κράτη-μέλη και ένα άλλο προέρχεται από το γεγονός ότι αυτά τα φάρμακα δεν συνταγογραφούνται ενώ επιπλέον κάπου υπάρχει και το πρόβλημα ότι τα φάρμακα αυτά επειδή προέρχονται από ορμόνες ε, δημιουργούν προβλήματα στο πόσιμο νερό. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά τα αντισυλληπτικά γίνονται lifestyle. Γι' αυτό υπάρχουν διαφορές στη συνταγογράφηση. Άλλοι γιατροί ανάλογα με τη χώρα συνταγογραφούν, αλλού γυναικολόγοι, αλλού παθολόγοι, αλλού δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι μπορείς να πας σε ένα φαρμακείο και να πάρεις ε, ε, σε, μετά από κάποια ηλικία αντισυλληπτικά χωρίς ε, συνταγή. Ούτε οι γυναικολόγοι, ούτε οι γιατροί λοιπόν εξετάζουν τους ασθενείς ούτε τους συμβουλεύουν τι να κάνουν και δεν τους συμβουλεύουν γιατί δεν τους θεωρούν ασθενείς, δεν τους θεωρούν ασθενείς, είναι κομμάτι της ζωής, έτσι, lifestyle. Θα έπρεπε λοιπόν να, χρησιμο... να, να συμβουλεύονται τον χρήστη. Δεν το κάνουν, εξού και οι παρενέργειες. Τώρα έχουμε και το πρόβλημα της κεντρικής ε, αδειοδότησης, το έθεσε η Ντάγμα, συμφωνώ μαζί της, και η φαρμακοεπαγρύπνηση. Είναι δύο τομείς που δεν έχουμε παρέμβει. Εμείς έχουμε την περίπτωση των κλινικών ελέγχων που, όπου η μετά τη χρήση συνέπεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα φάρμακα, τα, τα φάρμακα που χρησιμοποιεί ιδίως των, της τρίτης και τέταρτης γενιάς ε, έχουν πολύ μικρή ε, τεχνική, ε, κλινική εξέταση. Συχνά τα στοιχεία που βλέπουμε προέρχονται από τις φαρμακές εταιρείε. Όταν έχουμε επιστημονική έρευνα ανεξάρτητη βλέπουμε την αλήθεια. Σε πολλές περιπτώσεις οι κλινικές έρευνες δημοσιεύονται και εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ενώ πιστεύω ότι θα πρέπει η αίμα να το, παρουσιάζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, το πρόβλημα είναι και έλλειψη διαφάνειας. Το γαλλικό πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ε, ότι τα αντισυλληπτικά τρίτη και τέταρτη γενιά δεν μπαίνουν στην εθνική λίστα αποζημίωση των ιατρικών ω ιατρικά έξοδα. Αν δεν προχωρήσουμε σε αλλαγέ, θα συνεχίσουμε να έχουμε τα προβλήματα που σχολιάζουμε που τώρα, όχι στα αντισυλληπτικά αναγκαστικά, αλλά σε άλλα φάρμακα, με μη ανταγωνιστικέ ε, εμπορικέ πρακτικέ των φαρμακευτικών εταιριών που πολλέ φορέ δεν τηρούν τον νόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ακούσουμε και πάλι την άποψη των εμπειρογνωμών. Εγώ θα ήθελα να εμπλέξουμε πάλι και το θέμα της ευθύνης των ιατρών για προϊόντα όπως αναφέρθηκε προϊόντα lifestyle. Και ουσιαστικά πλήττονται ιδιαίτερα οι γυναίκες γιατί οι, οι άνδρες που παίρνουν τις αποφάσεις πολλές φορές δεν τους ενδιαφέρουν οι παρενέργειες για τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε λοιπόν να εμπλέξουμε τα πάντα πάνω στη γη, αλλά σίγουρα οι γιατροί έχουν πραγματικά μία ευθύνη για τα θέματα αυτά, δεν μπορούν να συνταγολογούν ε, αντισυλληπτικά ελαφρά την καρδία η για διαδικαστικό θέμα. Να ακούσουμε όμως εμπειρογνώμονες, όχι. Ναι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν μπορέσω να δώσω μία συνολική απάντηση χωρίς να σταθώ στα επιμέρους σχόλια. Πολλά από τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν τονίσει το γεγονός ότι εδώ δεν έχουμε ένα απλό θέμα. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα και θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη επισκόπηση οφέλους και κέρδους. Ξεκινάει πάντα από τον θεράποντα ιατρό ή από τον ε, γυναικολόγο που πρέπει να συζητήσει με, τον, με την ασθενή ποια είναι η καλύτερη θεραπεία ή η καλύτερη συνταγογράφηση. Τι γίνεται στη συνέχεια και πώς παρακολουθείτε αυτό αν υπάρχουν παρενέργειες. Να μην ξεχνάμε ότι η λεγόμενη αυθόρμητη αναφορά σημαίνει ότι εναπόκειται στους ε, ασθενείς και στους ιατρούς να εξασφαλίσουμε ότι η πληροφορία καταγράφεται και μεταφέρεται στις ανδρομόδιες αρχές. Εάν δεν υπάρξει μια αυθόρμητη παροχή πληροφοριών σε, για, τα, για τις παρενέργειες, δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Το ερώτημα τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε πέραν αυτών των ε, αυθορμήτων, των αυθορμήτων παροχών πληροφοριών. Έχουμε, ένα, έχουμε την πληροφορία από τις ε, φαρμακευτικές εταιρείες και σας λέω ότι εξετάσουμε και την δυνατότητα να κάνουμε μόνοι μας μελέτες που τελικά θα μας βοηθήσουν. Αυτό το οποίο τονίστηκε από την Κομισιόν είναι ότι τώρα έχουμε δεσμευτικά αποτελέσματα και για το Διάν και για τα αντισυλληπτικά συνδυασμένων ορμονών, ό,τι αποφασιστεί είναι δεσμευτικό για όλη την Ευρώπη. Θα είναι λοιπόν ακριβώς η ίδια, οι ίδιες οδηγίες χρήσεων. Αν αποφασιστεί αυτό θα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα τώρα του αν είμαστε αρκετά προορατικοί. Έχουμε από το Σεπτέμβριο του 2011 μια σύσταση από το Συμβούλιο για να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες στα φάρμακα. Υπήρξαν λοιπόν ε, μετατροπές <clears throat> και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση. Ένα κρατος μέλος το οποίο έχει την ευθύνη για τα προϊόντα τα οποία εγκρίνονται στο έδαφος του αποφάσισε να αναλάβει δράση και λόγω αυτού εμείς είμαστε εμπεπλεγμένοι και κάνουμε ό,τι μπορούμε το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε παροχή πληρών, πλήρους πληροφόρησης στους ιατρούς. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας επισκόψης θα ακούσουμε το δυνατόν περισσότερες απόψεις ασθενών και ιατρών που να ληφθούν υπόψη. Σας είπα ότι θα έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν συγκρούσεις συμφερόντων για αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων, αλλά επιπλέον από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και πάλι εκπροσώπους των ε, ε, ασθενών στην ΠΡΑΚ <clears throat> που θα μας δώσουν μια προσθέμενη αξία ώστε να ληφθεί πλήρως και η άποψή τους. Σας ευχαριστώ κύριε Βατών. Κυρία Ρέιν, σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ σε μερικά από αυτά τα συγκεκριμένα σημεία η κυρία Γκροστέτ αναφέρθηκε στο ότι πρέπει να ξέρουμε πολύ γρήγορα πού βρισκόμαστε. Και πρέπει να σας πω ότι με τις πληροφορίες που έχουμε για τα ενεργά συστατικά θα προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Ετέθη το ερώτημα γιατί θεωρούνται καλύτερα τα τρίτη και τέταρτη γενιά. Εμεί θα κοιτάξουμε όλα τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την ανεκτικότητα σε αυτά τα φάρμακα, για ορισμένε γυναίκε είναι πιο εύκολο να παίρνουν αυτά τα αντισυλληπτικά τρίτη και τέταρτη γενιά. Επίσης αναφέρεστε στην χρήση των φαρμάκων για, άλλες, για άλλους σκοπούς. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε καλύτερα με τη νέα μορφή οδηγιών χρήσεων. Άλλες χώρες έχουν ε, αναφέρει αντίστοιχα προβλήματα, ξέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν ξέρουμε για άλλες χώρες που έχουν τα ίδια προβλήματα όπως αυτά που έχουν ανακύψει στην Γαλλία, ώστε να μην υπάρχει ώστε να προτείνεται να μην χρησιμοποιηθεί πλέον το Διάν. Η κυρία Ρίβενς μίλησε για τα προβλήματα της φαρμακοεπαγρύπνησης και ακούσατε από τον κύριο πόσο μεγάλες προσπάθειες έχουν γίνει. Όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να βελτιώσουν την παροχή πληροφόρησης αλλά και να ενημερώσουν τους ασθενείς και να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της φαρμακοεπαγρύπνησης. Επίσης το θέμα της καλύτερης εκπαίδευση των του ιατρικού προσωπικού που είναι για μας μια τεράστια προτεραιότητα. Η κυρία Ρόσπαχ ρώτησε αν είχαμε στατιστικές για άλλους κινδύνους που θα μπορούσε να δώσει ένα γενικότερο πλαίσιο με τα στοιχεία που έχουμε για τα αντισυλληπτικά. Η κυρία Ροτ Μπέραντ ζήτησε μεγαλύτερη συνεκτικότητα και καλύτερη παροχή συμβουλών για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτό θα προκύψει από την επισκόπησή μας. Αναφέρθηκε επίση και το θέμα της ανεξαρτησία τη έρευνα. Η νέα νομοθεσία μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη χρησιμοποίηση των στοιχείων με τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου. Η συμπεριφορά των θεραπών των ιατρών είναι κάτι που πρέπει να μελετήσουμε επιπλέον και το θέμα της εμπορίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν θα το απολέσουμε από τον οφθαλμό μας. Το να, το θέμα της διαφήμισης και της πρόθεσης. Σε σχέση με τη χρήση των ε, ετικετών, ζητήσατε να ξέρετε για τη διαδικασία αυτή και αυτό ίσως μπορεί να το αντιμετωπίσει η Κομισιόν. Αναφερθήκαν επίσης τα θέματα της γενετικής για μια περαιτέρω μείωση του κινδύνου και αυτό θα είναι τμήμα της εξετασής μας. Τέλος, είναι χρήσιμο να σκεφτούμε τις μελέτες μετά από την έγκριση ενός φάρμακου, γιατί έχουμε με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να πάρουμε πιο ανεξάρτητα και πιο αξιόπιστα δεδομένα και ελπίζω ότι αυτή η επισκόπηση θα σας δώσει νέα στοιχεία για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προς όφελος όλων των γυναικών στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τη σύναψη και τις, και τις χρήσιμες απαντήσεις. Η Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Ναι, να απαντήσω σε κάποια θέματα που τέθηκαν προς την Επιτροπή. Προφανώς ε, η, η, δεν θα λύσουμε την αντιπαράθεση μεταξύ εθνικής άδεια και κοινοτική άδεια, ε, γιατί πρέπει να λειτουργήσουμε στο υφιστάμενο πλαίσιο. Όποιο μέτρο αποφασίζει σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφασίζεται βάσει του ελέγχου του κινδύνου. Εμείς θα πρέπει να το εφαρμόσουμε με, ένα, εναρμονισμένο τρόπο. Να υπάρχει δηλαδή εναρμονισμένη εφαρμογή ανεξάρτητα του τύπου ε, της άδεια. Προφανώς σε κάποιους τομείς θα πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι ευθύνη του κράτους μέλους. Φερπίνει αποφάσεις ε, για την τιμολόγηση. Αυτό είναι εθνικό θέμα υπό τον εθνικό έλεγχο. Πρακτική πρόθεση στην αγορά. Υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά εν τέλει η υλοποίηση του ελέγχου, η υλοποίηση και ο έλεγχος είναι εθνικές αρμοδιότητες. Οι αποφάσεις για το καθεστώς συνταγογράφησης των εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων, ναι, όταν υπάρξει ε, κεντρική αδειοδότηση θα συμφωνήσουμε επί ενός τρόπου συνταγογράφησης ή δε μη, τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν με τον α ή β τρόπο. Αυτή είναι η περιορισμοί του συστήματος το οποίο ζούμε. Αλλά το να μιλάμε για τρόπους νομοθεσίας για την ε, μορφή συνταγογράφησης και τις καλέ πρακτικές συνταγογράφησης είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Είναι σημαντικό νομίζω αυτό να το δούμε όχι ως ε, νομοθετικό αλλά ως ενημερωτικό στοιχείο. Δεν θα μπορούσα να σας δώσω λύση για το πώς θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε και να ελέγχουμε τις πρακτικές συνταγογράφησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άννα, ένα, ένα ερώτημα μονάχα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε προτείνω να μπει στην εμερήσια διάταξη μια ακρόαση, δημόσια ακρόαση για αυτό το θέμα, γιατί το θέμα παραμένει ανοιχτό. Μπορούμε λοιπόν να το συζητήσουμε παρετέρω στα πλαίσια μιας δημόσιας ακρόασης. Μερσή λοιπόν και νομίζω ότι οι συντονιστές θα πρέπει να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το θέμα αυτό. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εγώ έμαθα πολλά από αυτά που άκουσαμε. και είναι πολύ σημαντικό το ότι η Κομισιόν και ο Φορέας Φαρμάκων να αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας. Κλείνω τη συνεδρία. Σας υπενθυμίζω πάρτε όλα τα χαρτιά σας και θα ξεκινήσουμε στις 2.30 ε, και θα έχουμε να υποδεχτούμε τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρτε όλα τα χαρτιά σας μαζί σας.